Από τι φαίνεται, ο Επίτροπος ξέρετε κάπου έχει κολλήσει λόγω της απεργίας. Ας ξεκινήσουμε με ένα άλλο θέμα και όταν έρθει θα διακόψουμε τις διαδικασίες μας έτσι ώστε να συζητήσουμε μαζί του θα πρότεινα να περάσουμε στο σημείο 19 David Μάρτιν. Η πρόοδος... των τριμερών διαπραγματεύσεων. Θα δώσω το λόγο στον David Μάρτιν για να μας μιλήσει για την πρόοδο ή την έλλειψή της ε, για τον κανονισμό του πολιτού του δημοσιονομικού πλαισίου. Συγγνώμη, διόρθωνα πρόεδρος, για την πρόσβαση στην αγορά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για αυτή την ε, απρόσμενη τιμή. Η κατάσταση του κανονισμού είναι η εξή. Χθε είχαμε τον πρώτο τριμερή διάλογο Έχουμε τρία σύνολα τροποποιήσεων, τροπολογιών. Το πρώτο σύνολο έχει να κάνει με γλωσσικέ τροπολογίε, δεν υπάρχει πρόβλημα για το Κοινοβούλιο. Το δεύτερο σύνολο τροπολογιών έχει να κάνει με τι διατάξει περί όπου δεν σημειώσαμε ιδιαίτερη πρόοδο χτες αλλά ακούσαμε ότι υπάρχουν πρόοδοι στις διαπραγματεύσεις για τις συζητήσεις Omnibus 2 και φυσικά αν προχωρήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις ε, αυτό αφορά και συγκεκριμένα μέτρα για τον κανονισμό πρόσβαση στην αγορά και το κύριο θέμα αυτού του φακέλου είναι τα δεδομένα είναι η ημερομηνία, συγγνώμη, λήξης ε, του κανονισμού 1η ε, Ιανουαρίου 2014 από τη Μουσική Κομισιόν εννοεί το Κοινοβούλιο ψήφισε ε, για τον Ιανουάριο του 2016. Συζητήσαμε αυτό το θέμα χτες ε, και δεν σημειώθηκε περόδος, αλλά θέσαμε μία ημερομηνία την επόμενη εβδομάδα για έναν περαιτέρω τριμερή διάλογο και θα προσπαθήσουμε φυσικά ε, να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις αν και δεν ε, υπάρχει συμφωνία. Αρχίζουμε άτυπες διαπραγματεύσεις σήμερα με το Συμβούλιο για να δούμε αν μπορούμε να βρούμε συμβιβασμό. Πρόεδρος, όμως θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξη συμβιβασμού. Κοιτάξτε, είμαι σοσιαλιστής πάντοτε. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μάλλον όλοι συμφωνούν μαζί σας. Βλέπω ότι το ΕΛΚ συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό. Θα το δούμε για να είμαι ειλικρινής. Ε, κοιτάξτε, μεταξύ του 2014 και του 2016 υπάρχει και το 2015, αλλά δεν ξέρω ε, τι θα γίνει. Θα πρέπει να δούμε και αν το Συμβούλιο θα είναι προετοιμασμένο να υποχωρήσει. Μάλιστα. Συμφωνώ με την ανάλυση σας και εγώ περιβρισκόμουν εκεί και συμφωνώ Μπορούμε να διακόψουμε λοιπόν αυτό το σημείο εδώ. Let me welcome Να καλωσορίσω τον Επίτροπο Δεγκούκ. Ανυπομονούμε να τον ακούσουμε. Όπω γνωρίζετε, η τελική έκθεση τη κοινή ομάδα εργασία Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Ηνωμένων Πολιτειών δημοσιεύτηκε και συστήνει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια φιλόδοξη συμφωνία εμπορική συμφωνία και συμφωνία επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΠΑ. Ο Επίτροπος βρίσκεται εδώ για να μας παρουσιάσει την έκθεση αυτή και τι σημαίνει αυτή η πρωτοβουλία και να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Χωρίς χρονοτριβή θα του δώσω το λόγο γιατί έχουμε καθυστερήσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη γιατί καθυστέρησα. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν απεργίες των Βέλγων υπαλλήλων και έπρεπε να έρθω από το βόρειο τμήμα της πόλης ε, και ε, είχα προβλήματα. Όσον αφορά τώρα την ε, συνεργασία, ε, τη διατλαντική συνεργασία και το εμπόριο, είναι συνήθως ε, μια διατύπωση της οποίας γίνεται κατάγριση, χρησιμοποιείται για κάθε ευκαιρία, όμως σήμερα θα τη χρησιμοποιήσω σωστά. Πρόκειται να αρχίσουν οι μεγαλύτερες διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει ποτέ μεταξύ δύο πολύ μεγάλων οικονομικών ε, δυνάμεων. Ε, θα υπάρξει μεγαλύτερη ελεύθερη ζώνη, ζώνη ελευθέρου εμπορίου σε όλο τον κόσμο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για το διμερές εμπόριό μας και τις επενδύσεις μας στο μέλλον, αλλά και για την ανάπτυξη των κανόνων της Δόχα. Θα υπάρξει μεγάλος αντίκτυπος ε, στην ανάπτυξη και στις, στην απασχόληση κατέρωθεν του Ατλαντικού. Όταν θα αρχίσει λοιπόν να ισχύει αυτή η συμφωνία, ε, θα υπάρξει ενίσχυση κατά μισό της εκατό ε, το ΑΕΠ που σημαίνει δεκάδες ε, δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η αύξηση δηλαδή θα είναι περίπου τα δύο τρίτα του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό όταν προσπαθούμε να, να ανακάμψουμε από την, ε, από την κρίση και βέβαια είναι το φθηνότερο πακέτο ανάπτυξης και ενίσχυσης της οικονομίας ε, που μπορούμε να πετύχουμε. Χρειάζεται βέβαια πολιτική βούληση. Πρέπει να είναι συμβατοί όλοι οι κανόνες μας και να μειωθεί το κόστος ε, όταν αυτό είναι δυνατό και λογικό θα υπάρξουν λοιπόν συναλλαγές ε, για τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις, ε, μεταξύ των εταιριών, ε, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει και δέσμευση σε ανοιχτές αγορές και απελευθέρωση του εμπορίου, είναι δηλαδή το αντίθετο του προστατευτισμού. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι στρατηγικοί εταίροι που έχουν, έχουν την θέληση να κάνουν το βήμα για να συνεργαστούν και δεν είναι, δεν προκαλεί έκπληξη ότι το, οι ανακοινώσει ε, έτυχαν ιδιαίτερη υποστήριξη ε, σχεδόν ε, από όλους. Να σας μιλήσω για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να πω ότι να τονίσω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σήμερα να συζητήσω μαζί σας. Γνωριζόμαστε καλά και δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σημαντικό το Κοινοβούλιο και η συγκεκριμένη Επιτροπή είναι σημαντικά για μένα είναι ένας βασικός συνομιλητής για εμπορικά ζητήματα συμπεριλαμβανομένου βέβαια τη συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων δεδομένων ε, των διατυπώσεων ε, της ε, συμφωνίας φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν πολλές προτάσεις από πλευρά σας είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε αποτελεσματικό τρόπο οργάνωσης του συγκεκριμένου διαλόγου όπως επιθυμείτε κάποιοι μπορεί να είχαν αναρωτηθεί για τον τίτλο συμπορευόμαστε με τους ε, Αμερικάνους φίλους μας, ε, δεδομένου ότι η ομάδα υψηλού επίπεδου κατέληξε σε αυτήν την συμφωνία. Ε, θα μπορούσε να αποκληθεί διατλαντική συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων. Όμως πράγματι αφορά την, το εμπόριο και τις επενδύσεις και όταν βλέπω το ψήφισμά σας ε, του Οκτωβρίου του 2012 ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι με την τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών γιατί τα βασικά στοιχεία που είχατε αναφέρει έχουν συμπεριληφθεί. Περί τίνος πρόκειται λοιπόν. Ε, όταν μιλούμε για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Έχουμε δει την ε, τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου που, της οποίας προέδευσα εγώ μαζί με τον ε, Λον Κέρκ 14 μήνε σκληρή δουλειά. Αναγνωρίσαμε του τομεί που θα αποτελέσουν τμήμα των διαπραγματεύσεων, ε, όπω για παράδειγμα η δασβή, ε, τα υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά μέτρα, τα σχετικά ε, ζητήματα, τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, οι δημόσιε συμβάσει και εμπορικοί κανόνε, όπω για παράδειγμα οι πτυχέ που έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό. Φτάσαμε στο κοινό συμπέρασμα ότι μια περιεκτική συμφωνία που λαμβάνει υπόψη πολλά στοιχεία ε, εμπορίου και επενδύσεων, ε, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και ρυθμιστικών ζητημάτων, ε, θα είναι προς αμοιβαίο συμφέρον και των δύο. Επομένως, ε, οι πρόεδροι Ομπάμα, Μπαρόσο και Φανρόμπα ε, συμφώνησαν με την συμφωνία αυτή και είπαν ότι ε, είναι πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αρχίσει η διαδικασία, διαδικασία το συντομότερο δυνατόν και να αποστείλουμε τις σχετικές οδηγίες για διαπραγματεύσεις ε, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο τον επόμενο, την επόμενο μήνα. Δεν θα είναι κάτι εύκολο βέβαια η όλη αυτή ε, προσπάθεια. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε σε δύο χρόνια ε, την διαδικασία. Βέβαια είναι πιο σημαντικό να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους. Ε, αντί να μπούμε σε πολλές ε, λεπτομέρειες, καλύτερα να επικεντρωθούμε σε τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, πρέπει να απομακρυνθούν οποιαδήποτε δασμολογικά εμπόρια, εμπόδια συγγνώμη, και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να απελευθερώσουμε τομείς όπως τις δημόσιες συμβάσεις και την επένδυση, τις επενδύσεις. Έχουμε πολύ χαμηλούς δασμούς ούτως ή άλλως ήδη, κατά μέσο όρο 4% είναι οι δασμοί στις εισαγωγές μας. Ε, θέλουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με τους δασμούς τους, ε, και τα εμπόδια που βρίσκονται στο εσωτερικό των ε, κρατών, όπως για παράδειγμα η πιστοποίηση, κάτι το οποίο βέβαια είναι και χρονοβόρο και δαπανηρό. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε έτσι πολλά χρήματα, αλλά και να υπάρξει και μεγαλύτερη αξία για τους καταναλωτές μας και μεγαλύτερη επιλογή. Δηλαδή θέλουμε συχνά να καταργήσουμε ε, ε, δασμολογικά εμπόδια κατά 10% ώστε να μειωθεί και το κόστος προς τους καταναλωτές. Θέλουμε επίσης να βασιστούμε σε ε, παγκόσμια πρότυπα ε, για να υπάρξει ένα καλύτερο εμπορικό περιβάλλον κατά τα ερχόμενα χρόνια. Θα είναι δύσκολο βέβαια να το επιτύχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και ευχαρίστω να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Επίτροπε, για την σύντομη αλλά πολύ ουσιαστική παρουσίασή σας. Και τώρα τα μόνιμα μέλη η κυρία Γκότλιμπ από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, κύριε Επίτροπε. Και νομίζω πραγματικά ότι είμαστε πολύ ευτυχείς όλοι όταν ακούσαμε τον ε, πρόεδρο Ομπάμα, ο οποίος ε, δήλωσε ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι υπέρ της δημιουργίας αυτής της ε, μεγάλης ζώνης οικονομικής συνεργασίας. Σήμερα η συνεργασία μας με την άλλη όχθη του Ατλαντικού πρέπει σαφώς να τύχουν επεξεργασίας και αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ ευχάριστο. Το θέμα της Κίνας όμως, πόσο καιρό ακόμα θα διαρκέσει αυτή η διαπραγμάτευση. Έχετε εσείς ε, κάποιες ε, προθεσμίες, ημερομηνίες οι οποίες να σας φαίνονται ρεαλιστικές. Επίσης αυτή η συμφωνία για τις ελεύθερες συναλλαγές φυσικά έχει δημιουργήσει πάρα πολλές προσδοκίες. Αλλά θα ήθελα να ξέρω πόσο καιρό θα διαρκέσει. Ναι, περιμένουμε πολλά από το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων, αλλά υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι και κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε απογοήτευση αν δεν πετύχουμε αυτό που περιμένουμε και περιμένει ο περισσότερος κόσμος. Θα πρέπει λοιπόν ίσως να σκεφτούμε και μια εναλλακτική λύση, ένα άλλο σχέδιο, σε περίπτωση που υπάρχει μια σχετική απογοήτευση. Πώς μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την πρόοδο που ήδη έχει επιτευχθεί, εάν δεν προχωρήσουν όπως περιμένουμε οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σέτκε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, και εγώ θεωρώ ότι είναι μια ιστορική στιγμή, συμφωνώ μαζί σας και ότι υπάρχει πολιτική βούληση και από την Επιτροπή και από το Κοινοβουλίο. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και στήριξη της κοινή γνώμης. Εδώ βεβαίως θα πρέπει να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις και σε κριτική. Θα σας κάνω λοιπόν κάποιες δύσκολες ερωτήσεις. Η πνευματική ιδιοκτησία, και η άποψη της ομάδας υψηλού επίπεδου. Επίσης, το θέμα των αγροτικών προϊόντων. Έχετε σκεφτεί την εναλλακτική λύση να αποκλειστεί το θέμα της γεωργίας ή αυτό αποκλείεται κατά την άποψή σας. Επίσης βλέπετε τα επιμέρους ενδιαφέροντα και συμφέροντα, τα οποία ενδεχομένως κινδυνεύουν να θέσουν σε κίνδυνο το σύνολο της συμφωνίας. Επίσης, η άποψη των ε, Ηνωμένων ε, Πολιτειών, τα TPP, ποια είναι, αν θέλετε, η άποψη των ε, Ηνωμένων Πολιτειών ποια είναι η άποψη των πολιτιών σε σχέση παραδείγματος χάρη με το Ομοσπονδιακό Αμερικανικό κράτος. Ξέρουμε ότι εδώ υπάρχουν ρήτρε των επιμέρους πολιτιών όπως παραδείγματος χάρη της ε, πολιτείας της Πενσιλβάνια ή άλλων πολιτιών. Εμείς ε, θα θέλαμε να μην διακοπήσει η επικοινωνία μεταξύ μας και να συνεργαστούμε στενά έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και την στήριξη της κοινή γνώμης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στέρντι, ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε, είναι εξαιρετικό αν θέλετε, το καλύτερο, το πιο θετικό μήνυμα που ακούσαμε εδώ στην Επιτροπή μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σας συγχαίρω λοιπόν πάρα πολύ για το ότι έχετε πετύσει μέχρι τώρα. Θα ήθελα να πω ακριβώς αυτό που είπε και η κυρία Σάλκε. Εγώ έχω συζητήσει με πολλούς από τις Ηνωμένε Πολιτείε για τα θέματα της γεωργίας. Το θέμα είναι ότι όλοι θεωρούν ότι πρέπει να συμπεριληφθούν τα θέματα αυτά στην διαπραγμάτευση. Την άλλη μεριά έχουμε την ΚΑΠ. Μήπως ε, οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι ευκαιρία να ξεφορτωθούμε την ΚΑΠ. Ε, εγώ προσωπικά θα το πρότεινα. Αλλά σκεφτείτε πραγματικά ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μεγάλη δυσκολία στα πλαίσια των διαπραγματεύσεών μας. με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Ξέρω εδώ ότι ξεπερνάω κατά κάποιο τρόπο τις θερμοδιατές και το, αυτό που θα έλεγα, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα των των ε, γενετικά τροποποιημένων ε, καλλιεργειών και το θέμα των εισαγωγών. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση το θέμα αυτό το συγκεκριμένο το, της Γεωργίας να καταστρέψει όλη μας τη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Ζαμπού. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι ο Ρόμπερ Στουαρντή θα ήταν ο καλύτερος, αν θέλετε, εταίρος και εκπρόσωπος για να προχωρήσουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να μην ολοκληρωθούν ποτέ. Εγώ είμαι υπέρ του να δημιουργήσουμε μια κοινή θέση και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Ευρώπη και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και υπάρχει κάτι που ακόμα με εντυπωσιάζει. Όπως είπατε, μιλάμε για το 0,5% ανάπτυξης. Είπατε ότι αυτό ε, περιέχει η πρότασή σας. Και ουσιαστικά αυτό θα καταλήξει σε 2% αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Αν είχαμε ακούσει όλες τις προηγούμενες προτάσεις που περιέχονται σε όλες τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει από το 1994 μέχρι σήμερα και αν κάθε φορά είχαμε υιοθετήσει μείωση των δαπανών, λιτότητα και φιλελευθεροποίηση των υπηρεσιών και είχαμε όντως όλη αυτή την επιπλέον ανάπτυξη που μας είχαν υποσχεθεί θα ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση από ότι είναι η Κίνα σήμερα και θα είχαμε περισσότερες νέες θέσεις απασχόλησης από οποιοδήποτε άλλος μέρος του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει αστείευομαι και οι υπηρεσίες που κάνουν την μελέτη αντικτύπου ίσως θα έπρεπε να αξιολογήσουν τις υποσχέσεις αυτής της διαπραγμάτευσης. Γιατί μοσνήμως μας λένε αν υπογραφεί αυτή η συμφωνία θα έχουμε 1% ή 0,5% ε, επιπλέον ανάπτυξη και τόσες θέσεις απασχόλησης. Και μετά υπογράφουμε τη συμφωνία και δεν βγαίνει τίποτα από όλα αυτά αληθινό. Αν δείτε την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας σήμερα, θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι όλα αυτά δεν υλοποιούνται και δεν έχουν καμία βάση. Επί τους ουσίας τώρα θα χρειαστείτε σαφώς την υποστήριξη και την εντολή του Συμβουλίου, όπως ακριβώς και ο πρόεδρος Ομπάμα χρειάζεται την στήριξη και την εντολή του Κογκρέσου. Μπορείτε να μας πείτε πώς έχει η κατάσταση στο Κογκρέσο όσον αφορά τις διάφορες πτυχές, γιατί ο Ρόμπερτ έχει δίκιο. Για την ΚΑΠ θέλουν να συμπεριληφθεί. Έχει δίκιο. Θέλουν επίσης οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί επίσης να συμπεριλαμβάνονται. Επίσης τα δικαιώματα των επενδυτών. Ξέρουμε σήμερα ότι πρέπει να ενισχυθούν οι επενδυτές, είτε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα ενημέρωσης των πολιτών, της ομάδας των πολιτών και να δούμε πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι μεγάλοι επενδυτές και οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας. Είδατε το σκάνδαλο, το οποίο δεν είναι σήμερα υγειονομικό σκάνδαλο, με το κρέας των αλόγων. Πρόκειται όμως για ένα φαινόμενο που οφείλεται καθαρά στην παγκοσμιοποίηση. Σήμερα βλέπουμε τους Ευρωπαίους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε μια πολύ δεινή κατάσταση και την ίδια ώρα ενώ υπάρχουν τόσες εξαγωγές προς το Περού, προς ε, άλλες τρίτες χώρες οι οποίες θα μπορούσαν να τους δώσουν κάποιες δυνατότητες, εμείς να βρισκόμαστε σε αυτήν την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και πέρα από τις υποσχέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την επιπλέον ανάπτυξη, θα πρέπει εδώ να ξαναδούμε το πώς η ευελιξία μας ζητούν όσον αφορά τα πρότυπα που υιοθετούμε και εφαρμόζουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. το θέμα της ανταγωνιστικότητας που είναι ένα σημαντικό θέμα σε όλες μας τις χώρες. Αυτή η ανταγωνιστικότητα πώς θα ενισχυθεί. Θα ενισχυθεί μέσω της μείωσης των δαπανών είτε θα ενισχυθεί μόνο μέσω της ε, νέας, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας. Και αυτό βεβαίως θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται από κανόνες αυστηρότερους κοινωνικούς περιβαλλοντολογικούς. Είμαστε λοιπόν ναι υπέρ της ενίσχυσης του εμπορίου, υπέρ της διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά για τη ρύθμιση και όχι για την απελευθέρωση του εμπορίου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά τον προηγούμενο μιλτή και συμφωνώ. Καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε σε μία εφορία και θα πρέπει αν θέλετε να ξαναδούμε λίγο την ιστορία αυτών των διαπραγματεύσεων και να δούμε ότι έχουμε περάσει και από πολλές παρόμοιες φάσεις. Θα ήθελα να πω Όσον αφορά τα TTIP και την διμερή εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτεών θα πρέπει να δούμε και τα πολιτιστικά και όλες τις άλλες πτυχές που συμπεριλαμβάνονται. Και κατά την απόψη μου, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν σοβαρές διαφορές νομοθεσίας. Και σήμερα Ακούσατε τα πορίσματα και τις προτάσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου. Αλλά ακριβώς επειδή υπάρχουν σοβαρές διαφορές στην νομοθεσία, επειδή υπάρχουν σοβαρές διαφορές προσέγγισης, νοοτροπίας, όσον αφορά τα δικαιώματα ενημέρωσης των πολιτών, παραδείγματο χάρη. Και αυτό δεν είναι ένα καθαρά εμπορικό θέμα, είναι κάτι που διέπει γενικότερα τις σχέσεις μας. Πώς λοιπόν εμείς μπορούμε σήμερα να ξαναδούμε αυτές τις διαπραγματεύσεις συμπεριλαμβάνοντας και όλες αυτές τις πτυχές. Πώς δηλαδή οι αρμόδιοι επίτροποι, προχωρούν σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις στις διάφορες υπηρεσίες και τομείς αρμοδιότητας των Επιτρόπων στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς οραματίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συνέχιση αυτών των διαπραγματεύσεων συμπεριλαμβανομένων και όλων αυτών των ε, επιμέρους τομέων. Δεύτερον, σήμερα μιλούμε για μια διαπραγμάτευση που θα καταλήξει ενδεχομένως σε μια συμφωνία η οποία θα πρέπει να είναι προς όφελος των πολιτών. Ανάπτυξη, περισσότερη απασχόληση και αυτό σαφώς δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί αυτό το χρόνο, αλλά θα προχωρήσει και στην επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν πραγματικά το ερώτημα που θέτει ο Αμερικάνος ε, καταναλωτής, ο Αμερικάνος πολίτης. Τι θα μου αποφέρει εμένα αυτή η συμφωνία, να το θέσουμε και εμείς. Και εδώ στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, θα πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα λέγοντας ναι αυτή η συμφωνία θα επηρεάσει θετικά τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Επαναλαμβάνω, με περισσότερη ανάπτυξη, με περισσότερες θέσεις απασχόλησης και η κοινοτική μέθοδος εδώ θα πρέπει ίσως να αξιολογηθεί και να δούμε αν θα πρέπει να διατηρηθεί ή αν θα πρέπει να αλλοιωθεί. Σήμερα ε, μιλάμε για μια διαπραγμάτευση στην οποία συμπεριλαμβάνονται 27 κράτη-μέλη. Έχετε σήμερα κάποιες ενδείξεις όσον αφορά αυτές τις πολυμερείς ε, συμφωνίες. Εμείς, παραδείγματος χάρη, χθες μιλήσαμε για τις ε, δημόσιες ε, συμβάσεις, δημόσιες προμήθειες. Ένα τέτοιο θέμα θα πρέπει σαφώς να αντιμετωπιστεί και τον προτέρων, να προετοιμαστεί. Όντως υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές στην νομοθεσία. Διαφορές και αναρωτιέμαι αν υπάρχει μία ομάδα διαπραγματευτική η οποία να προετοιμάζει όλα αυτά τα θέματα γιατί πραγματικά εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα και θα θέλαμε να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια ομάδα η οποία προετοιμάζει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εδώ ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύριο ερωτήσεων. Τώρα έχω ένα πρόβλημα. Συνήθως ε, έχουμε τις ψηφοφορίες αυτή την ώρα. Αλλά βλέπω ότι ζητούν ε, και άλλοι το λόγο για το δεύτερο γύρο. Θα πρότεινα λοιπόν να δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Κατόπιν ε, να διακόψουμε για την ψηφοφορία και θα συνεχίσουμε για το δεύτερο γύρο και για τις τελικές παρατηρήσεις του Επιτρόπου. Συμφωνείτε? Ας δώσουμε λοιπόν το λόγο στον Επιτρόπο για να απαντήσει στον ε, πρώτο γύρο για να υπάρχει αμεσότητα στις απαντήσεις και κατόπιν θα διακόψουμε για την ψηφοφορία και θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο ερωταπαντήσεων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Πίτρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, πρέπει να ζητήσουμε τώρα εντολή από το Συμβούλιο. Είναι σχεδόν έτοιμη θα καταθέσουμε τις επόμενες ε, εβδομάδες, αρχές Μαρτίου. Συνήθως χρειάζονται τρεις μήνες ε, για τη συζήτηση αυτή στο Συμβούλιο. Έχουμε κατά νου να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή το αργότερο στο Συμβούλιο των Υπουργών Εμπορίου. Νομίζω στις 13-14 Ιουνίου είναι το Συμβούλιο. Ιδανικά θα ήταν νωρίτερα. Γιατί μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ακόμη και στην TPC, σε οποιαδήποτε σύνθεση δηλαδή. Αυτή είναι η προθεσμία λοιπόν που έχουμε κατά νου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, τώρα αυτή πρέπει να... Ο πρόεδρος πρέπει να το κοινοποιήσει το Κογκρέσο και υπάρχει μια περίοδο, περίοδος 90 ημερών, στη διάρκεια της οποίας μπορεί να κάνει παρατηρήσεις στο Κογκρέσο. Δεν ε, υπάρχει διαδικασία fast track στις ΗΠΑ και δεν ξέρω αν θα ζητήσουν τέτοια διαδικασία γιατί τη χρειάζονται όχι μόνο για αυτή τη συμφωνία και για αλλά και για την TPP. Όμως τώρα έχουμε αυτή την περίοδο 90 ημερών και αυτό σημαίνει ότι θα είναι δυνατόν επίσημα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα, που θα λάβει χώρα περί τα μέσα Ιουνίου. Αυτό έχουμε κατά νου λοιπόν. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν εργαζόμαστε ήδη για την τεχνική προετοιμασία όλων αυτών. και ήδη το κάναμε αυτό και κατά τη σύνταξη της έκθεσης, γιατί υπήρξαν, υπάρχουν αρκετά τεχνικά ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε. Δηλαδή, τι θα κάνουμε με το πρόβλημα των προτύπων και της προσέγγισης. Συνεχίζουμε λοιπόν να εργαζόμαστε από αυτού, αλλά επίσημα θα ξεκινήσει η διαδικασία μέση Ιουνίου. Ιδανικά εκτός και αν πει έχει το Συμβούλιο. Όπως φαίνεται να αναμένει ο κύριο Ζαντό. Μεγάλες προσδοκίες. Δεν ξέρω. Προσπάθησα να είμαι ρεαλιστικός. Νομίζω ότι είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τις ε, κάνουμε και αν καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία θα είναι καλό και για τις δύο οικονομίες μας ε, και για την Ευρώπη και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, και για τη γεωστρατηγική μας θέση. Υπάρχει τώρα η βούληση να τα δοκιμάσουμε. Αυτή η βούληση δεν υπήρχε για αρκετό καιρό. Ξέρετε ότι η Μερκεμόρ πριν 6 χρόνια το προσπάθησε για πρώτη φορά και το αποτέλεσμα ήταν κάποιες επιτυχίες στο Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο και αυτό συνέβαλε στην βούληση και στην ελπίδα να προσπαθήσουμε να έχουμε τέτοιες πλήρεις συμφωνίες όμως ε, δεν ε, υποτιμώ τα προβλήματα που υπάρχουν και από τις δύο προβλές υπάρχει τώρα σχέδιο Β, όχι. Τελειώνει η δική μου θητεία, σε ένα μισό χρόνο δεν βλέπω την αναγκαιότητα να έχω τέτοιο σχέδιο Β, εναλλακτικό σχέδιο. Και δεν με ενδιαφέρουν και τόσο αυτά τα εναλλακτικά σχέδια. Προτιμώ να χάνω. Will you develop Uh, Θα αναπτύξετε κάποιο. Δηλαδή προπαθείτε, προτιμάτε την ε, πλήρη αποτυχία από ότι ένα μερικό αποτέλεσμα. Λέτε ναι, μάλιστα. Όταν έχει κανείς τον ελεκτικό σχέδιο δεν πρέπει ποτέ να το πει. Ναι, είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε δημόσια υποστήριξη. Για όλα αυτά χρειαζόμαστε καταρχήν υποστήριξη από το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Αλλά διαφάνει πρόσφατα ότι χρειάζεται και δημόσια υποστήριξη και σε αυτά τα πολύ δύσκολα θέματα, όπως είναι τα δικαιώματα των διανοητικής η Γεωργία. Να ξεκινήσω με τη Γεωργία. Υπήρχαν πολλές ερωτήσεις ε, γι' αυτό θα είναι τμήμα των διαπραγματεύσεων η Γεωργία. Και για να είμαι ειλικρινή, η Γεωργία θα είναι σημαντικό τμήμα των διαπραγματεύσεων. Αλλά θέλω επίση να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται να θέσουμε επιτάπητος εφιστάμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δούμε το παράδειγμα των ε, γενικά τροπημένων οργανισμών, υπάρχει νομοθεσία για το θέμα αυτό που καθεστά δυνατόν να υπάρχει καταγραφή των γενικά τροπημένων οργανισμών και υπάρχει πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2010 σύμφωνα με την οποία θα αλλάξει το καθεστώς ε, για την καλλιέργεια. Αργαζόμαστε στα πλαίσια της εφιστάμενης νομοθεσίας ή στα πλαίσια της νομοθεσίας που έχει ήδη υιοθετηθεί. Και δεν μπορεί να αλλάξει κανείς τη νομοθεσία μέσω μια συνθήκη, να είμαστε ξεκάθαροι από αυτό. Και το ξέρουν και οι Αμερικανοί. Από την άλλη, δεν βλέπω γιατί θα έπρεπε να φοβόμαστε τόσο τη Γεωργία. Γιατί είναι αλήθεια ότι σε ένα βαθμό εξακολουθούμε να προστατεύουμε τη γεωργία μας, το ίδιο κάνουν και οι Αμερικανοί. Και ακόμη περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μερικές φορές είμαστε και οι δύο σε γκρίζα ζώνη. Δεν ε, καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να φοβόμαστε τόσο να το συζητούμε αυτό λες και θα επρόκειτο για το τέλος της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής. Κάτι που ζήτησε ρητά και ο κύριος Στέρντι. Ναι, ναι, μου αρέσουν τα άκρα για να μπορέσω να καταλήξω σε συμβιβασμό για το IPR, την πνευματική διοκτησία. Θα υπάρχει και ένα κεφάλαιο σχετικά στη συμφωνία. Το προωθούμε. Και επειδή θα υπάρχει μια συζήτηση και για τι γεωγραφικέ ενδείξεις ε, που εντάσσεται στη συζήτηση για τα, για τα δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα θέματα θα εμφανιστούν για τους γεωγραφικούς δείκτες και αυτοί τους προστατεύουν, αλλά με άλλο τρόπο, μέσω εμπορικών σημάτων που είναι ιδιοκτησία εταιριών μέσω ειδικών χαρακτηριστικών γεωγραφικών δικτών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών ε, σημειώσαμε τεράστια πρόοδο σε αυτό το θέμα. Δείτε τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κεφάλαιο για τις γεωγραφικές ενδείξεις και με την Κολομβία και με τον Καναδά. Επομένως, σημειώνουμε πρόοδο με το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων και θέλουμε να τη συζητήσουμε και με τους Αμερικανούς. Δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με αυτό. Προσπαθήσατε να κάνετε μία έμεση αναφορά στην άκτα. Είναι ένα δύσκολο σημείο αυτό. Δεν πρόκειται να ξανανοίξω αυτή τη συζήτηση, ειλικρινά. Δεν είμαι μεζοχιστής Αν ε, η Κομισιόν ε, προωθήσει νέα βασική νομοθεσία που νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνει, τότε θα ξαναδούμε το ζήτημα αλλά τώρα δεν πρόκειται να το κάνω από την πίσω πόρτα. Ο σύνδεσμος στην TPP. Αυτές είναι ξεχωριστές διαπραγματεύσεις και βλέπετε ότι είναι, έχουμε μια εταιρική, διατλαντική εταιρική σχέση, σχέση επενδύσεων βλέπετε ότι μιλάμε για εμπόριο και επενδύσεις. Το λέει και το όνομα της συνθήκης. Η TPP είναι ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εγώ πιστεύω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα έχουν μια καλύτερη δυνατότητα να υλοποιήσουν την TPP αν καταρχήν συμφωνήσουν με τους Ευρωπαίους γιατί η συμφωνία με τους Ευρωπαίους θα είναι μια συνθήκη σφαιρική και σε βάθος και η TPP θα είναι πολύ πιο δύσκολο να υλοποιηθεί αν δεν υπάρχει και το πρώτερο συμφωνία μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η προσωπική μου εντύπωση. Βέβαια θα είναι δικό μου πρόβλημα τελικά. Λοιπόν, ε, τώρα για τις προμήθειες σε κρατικό επίπεδο δεν είναι κάτι καινούργιο. Ισχύει και με τον Καναδά και με την Ινδία. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Φυσικά το Buy American δεν πρέπει να αντικατασταθεί με το Buy South Dakota. Αγοράστε από την Νότια Dakota. Και το Buy American δεν ανήκει σε μια τέτοια εταιρική σχέση εμπορική και επενδύσεων. Φυσικά θα πρέπει να συζητηθεί πλήρω γιατί θα ήταν εντελώ αντίθετο στο πνεύμα και στο περιεχόμενο μια τέτοια συμφωνία, κύριε Στάρτη. δεν ε, θα ξεφορτωθούμε την κοινή αγροτική πολιτική και οι γενετικά τροποποιημένες ε, καλλιέργειες είναι κάτι φυστάμενο. Κυρία Ζαντό, καταρχήν για τα ποσοστά. Εμένα δεν μου αρέσουν ε, τόσο τα ποσοστά, αλλά κάναμε μία μελέτη, δεν είμαστε εμείς η Κομισιόν που έκανε τη μελέτη αυτή πριν από την ε, έναρξη των διαπραγματεύσεων έγινε μια μελέτη αντικτύπου από ένα οργανισμό ε, και έφτασαν ε, στην εκτίμηση του 0,5 έως 1% μα, μα, βραχυπρόθεσμα και στο 2% μασοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Κατόπιν με όλες τις συμφωνίες από το 1996 αναφερθήκατε στις συμφωνίες αυτές. Ε, κοιτάξτε, εγώ είμαι αρμόδιος για αυτή τη θέση από το 2010. Είμαι πεσμένο ότι αν ε, δεν βρισκόμαστε σε βαθιά κρίση αυτή τη στιγμή είναι χάρη στο εμπόριο. Και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε ανά φάκελο και ανά χώρα. Ξέρετε ότι η Ιταλία λόγου χάρη είναι η πρώτη φορά από το 1999 που σημείωσε αύξηση εξαγωγών στα πλαίσια του εμπορίου. Η Ισπανία κάνει πρόοδος. Εξάγει περισσότερο προς τον ίδιο κόσμο, όχι προς τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα μπορούσαμε να το δούμε όλα αυτά λεπτομερώς χάρη στο εμπόριο δεν βρισκόμαστε σε βαθιά κρίση. Και αν πράγματι πιστεύετε ότι ε, μπορούμε να αποκαταστήσουμε αυτό στον φιλοφερθήκατε, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, γιατί οι άνθρωποι προέβαιναν σε εμπορικές συναλλαγές από τις απαρχές του είδους. Πάντα αυτό έκαναν. Δεν υπάρχει λόγος ξαφνικά να διακόψουν κάτι τέτοιο. Και κατόπιν αν δούμε το εμπορικό ισοζύγιο, αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κέρδη. και έχουμε όφελος. Υπάρχει θετικό εμπορικό ισοζύγιο. αγαθά, υπηρεσίες ε, και η γεωργία όλα μαζί φτάνουν περίπου στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ και τα χρειαζόμαστε όλα γιατί έχουμε το ίδιο έλλειμμα για το ρηκτό και την ενέργεια. Και τελικά πρόκειται για ένα δεδομένο. Γιατί αν ε, δεν υπάρχει χρυσό στο επέδαφο, δεν μπορεί κάποιο ε, να ε, πάει να το βρει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή η ιδέα περί αυτάρκειας δεν υπάρχει. Και είστε πολύ ευφύς για να μην το γνωρίζετε. Ο κ. Ζαντώ, δεν θα, θα με κάνετε να αλλάξει γνώμη με τα κοπλιμέντα σας. Εδώ δεν μιλάμε για το εμπόριο, μιλάμε για το περιεχόμενο της συμφωνίας, μάλιστα. Σας ευχαριστώ για τη μικρή παρέκκληση. Αναφέρθηκε στο παράδειγμα του κρέατος αλόγου. Από όσο γνωρίζω, αυτό που συμβαίνει τώρα δεν έχει καμία σχέση με την παγκοσμιοποίηση. Φαίνεται να προέρχεται το κρέας αυτό από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ε, και άτιμοι έμποροι και στη Γαλλία. Και σε ένα στάδιο από παγκοσμιοποίηση στη Γαλλία. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στη Γαλλία που εξαπατούν. Κύριε Σόλτς. Νομίζω ότι δίκιο έχετε. Όταν λέτε ότι υπάρχουν τεράστιες πολιτισμικές διαφορές. Γιατί συνεχώ μιλάμε για τεχνικά, τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο, εσωτερικού φραγμούς, αλλά ξέρετε ότι πολλέ φορέ ε, υπάρχουν πολιτιστικέ διαφορές. Και πιστεύω ότι θα είναι το πιο δύσκολο να ξεπεράσουμε αυτές τις πολιτιστικέ διαφορές. Θα βρούμε κοινό έδαφο για να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να λάβουμε υπόψη και ναι, θα συνεχίσουμε με το Διατλητικό Οικονομικό Συμβούλιο και τις διάφορες συζητήσεις εκεί. Έχουμε, τους χάρη, το Secure Traders, τους ασφαλίτες εμπόρους, ε, δηλαδή όταν ελέγχεται ένα εμπορευματοκιβώτιο στην Ευρώπη δεν χρειάζεται να ξαναελεγχθεί στις ΗΠΑ Και έχουμε προτάσεις από πάρα πολλούς κλάδους, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην TPIP και εν μέρει αυτό είναι το αποτέλεσμα όσων είχαμε συζητήσει στο Συμβούλιο στο παρελθόν. Και η τελευταία σας ερώτηση. Αν αυτό θα βοηθήσει την εκβιομηχάνηση της Ευρώπης. Νομίζω ότι η εκβιομηχάνηση της Ευρώπης εξαρτάται για το αν ε, μπορεί να γίνει μεγάλη πρόοδος στην καινοτομία και στην παραγωγή. Αν ε, πρέπει να ανταγωνιστούμε με την Ινδία και την Κίνα για, και με τη Βραζιλία για την αύξηση παραγωγής, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες ειδικέ αγορές που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εκ νέου και θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα στην παραγωγή αγαθών που έχουν ένα παράγοντα εγκύτητας. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό μπορούμε να μιλάμε για νέα εκβιομηχάνηση, αλλά για να έχουμε μια καλύτερη ιδέα γι' αυτό και πρόκειται για μια εντελώ διαφορετική συζήτηση, δεν πρέπει να έχουμε κατά νου τι βιομηχανίε και του κλάδου του παρελθόντο, αλλά του μέλλοντος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε πίτροπε. Θα διακόψουμε λιγάκι εδώ τη συζήτησή μας για να περάσουμε στην ε, ψηφοφορία. Αν θέλετε μείνετε μαζί μας ή αν θέλετε για 15 λεπτά μπορείτε να πιείτε έναν καφέ. Δεν μπορούμε να σας το σερβίρουμε όμως ε, σήμερα τον καφέ. Είναι εκεί ο καφές και μπορείτε να πάτε να πάρετε μόνοι σας. Okay. Thank you.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 Παρακαλώ καθίστε, καθίστε. Πρέπει να έχουμε ησυχία στην αίθουσα για να κάνουμε την ψηφοφορία μας. Παρακαλώ πολύ μην συζητάτε μέσα στην αίθουσα. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 14. Εμπόριο και ανάπτυξη βασισμένη στις επενδύσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Έκθεση Τόκια Σαΐφη. Να αρχίσουμε με τη συμβιβαστική 140 τροπολογίες, αλλά υπάρχουν πολλές συμβιβαστικές, οπότε μην ανησυχείτε. Λοιπόν, ας περάσουμε λοιπόν. Συμβιβαστική τροπολογία παριθμών 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 41 λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεβε 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμπεβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμπεβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμπεβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 65. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 66. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 67. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος της 67. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται όντως. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ καταπίπτει 106 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΔΕΒΕ 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΔΕΒΕ 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ντεβε 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ντεβε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, διορθώνει ο πρόεδρος. 120 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 132 και 140 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεβε 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 100... 136, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος του δεύτερου τμήμα της 136. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Δε 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΔΕΒΕ 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έλεγχο ζητάτε. Καλά. Εντάξει. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας το είπα. Μπορείτε να με πιστεύεστε. Αιτιολογικές σκέψεις. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Τροπολογία 12 υπέρ. Καταπίπτει, λέει ο πρόεδρο. Συμβιβαστική 2 λοιπόν υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά απόχέ. απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά α, α, εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όλες μαζί τις, ψηφοφο... τις... τις τροπολογίες από την 4 μέχρι τη 10. Τις ψηφίζουμε όλες μαζί. 4 έως 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ υπέρ. Υπάρχει κανένας, κανένας που διαφωνεί. Όχι. Οπότε ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικός. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία, 23 ψήφοι υπέρ και μία ψήφος κατά και τρεις αποχές. Συγχαρητήρια, Τόκια Σαΐφη. Περνάμε στη δεύτερη και τελευταία μας ψηφοφορία για σήμερα. Γιάννικ Ζαντού είναι ο εισηγητής μας. Γνωμοδότηση προς την Ήτρε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας. Συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τότε γιατί χρειαζόμασταν ε, δύο τμήματα στην ψηφοφορία. Τροπολογία 10 υπέρ Α, καταπίπτει, καταπίπτει. Καταπίπτει. Πάμε στη 15, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κύριε Φιέλνερ, 18 υπέρ, κατά, αποχές, 18, 18 λέει ο πρόεδρος, 18. Πάλι Φιέλνερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Ξεχάσαμε τη συμβιβαστική τρία, λέει ο πρόεδρος. Τι ψηφίζουμε τώρα. Ήθελα να πάω πιο γρήγορα, αλλά... Τρία λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 καταπίπτει. Τι ωραία. Για τον κύριο Φιέλνερ καλό αυτό. 29 υπέρ. Α, κατά τμήματα, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Το πρώτο τμήμα καταπίπτει. Άρα ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Ωραία. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Να ρωτήσω πρώτα αν διαφωνεί κανείς. Με την προφορική τροπολογία 1. Όχι, ωραία, ψηφίζουμε τότε. Προφορική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικώς γιατί δεν είμαι σίγουρος. Για την προφορική τροπολογία ένα μιλάω. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε ότι εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία, γι' αυτό να σηκώνετε καλά τα χέρια. Τουλάχιστον οι ηγέτες, γιατί εγώ πάντοτε τους ηγέτες ακολουθώ. είναι πιο εύκολο να καταλάβει κανεί το αποτέλεσμα. Συγγνώμη, ζητώ προς του υπόλοιπους συναδέλφου. Αν υπάρχουν αντιφρονούντες δεν τους λάβω υπόψη, παρά το γεγονός ότι είμαι και εγώ καμιά φορά αντιφρονών. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχο ζητάτε. Τις 24, τις 34, συγγνώμη, υπέρ Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές επαναλαμβάνω συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι να ελέγξουμε καλώς άρχεται η ψηφοφορία And what is... πέρασε απορρίπτεται Υπήρχαν αντιφρονούντες αυτή τη φορά. 37 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται αυτή τη φορά κύριε Φιέλνερ, συγχαρητήρια Συγχαίρω το συγκεκριμένο συνάδελφο που υπέβαλε αυτή την τροπολογία. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικός, έναρξη. And Πέρας. 24 υπέρ, ένας κατά, τρεις αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Ζαντού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Okay, let's come back to... Επανερχόμαστε λοιπόν στη συζήτηση που έχουμε με τον Επίτροπο Ντεγκούχτ, δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Αν θέλετε να βγείτε από την αίθουσα παρακαλώ πολύ σύντομα και με ησυχία να το κάνετε. Βλέπω ότι υπάρχουν πολλές συζητήσεις στο πίσω μέρος της αίθουσας. Okay, second round. Δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Θα αναγκαστώ να περιορίσω τον αριθμό των ομιλητών. Χρόνος ομιλίας τρία λεπτά. Σάιμον από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε να σας υπενθυμίσω, δεν ανήκω στο ΕΛΚ από το 2009. Με θέλουν να γυρίσω, αλλά εγώ δεν έρχομαι. Είμαι πολύ ευτυχής στην ομάδα που βρίσκομαι σήμερα. Να να χαίρομαι που εκτιμάτε το χιούμορ μου. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να αναφερθώ σε κάποια από αυτά που ήδη συζητήσαμε, το οποίο όμως είναι στρατηγική σημασίας. Παραδείγματο χάρη, όσον αφορά την διαπραγμάτευση, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εμείς πιέζουμε τη Σιγκαπούρη για ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης. Από την άλλη μεριά στο εσωτερικό αυτής της συμφωνίας ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε, ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί πιέζουν πάρα πολύ για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Πώς αυτά τα δύσκολα θέματα θα τα ξεπεράσετε, πώς ε, σκέφτεστε να το κάνετε, περιμένετε να προκύψουν οι δυσκολίες ή θα προετοιμάσετε το έδαφος με κάποιες κινήσεις. Ξέρω ότι είστε πολύ ειλικρινείς και πάρα πολύ ε, συγκεκριμένως ε, όσον αφορά την, το χρονοδιάγραμμα το ευρωπαϊκό. Πώς ε, έχει όμως το χρονοδιάγραμμα από μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών σκέφτονται να γίνει ένας και ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων. Ξέρω ότι έχουμε τις εκλογές, άρα υπάρχει και η δεύτερη εντολή και ο επίτροπος για εμπορικά θέματα που ενδεχομένως θα σας ε, ε, αντικαταστήσει. Ο κύριος ε, Ζαντό έθιξε κάποια από αυτά τα θέματα. Ξέρω ότι πολλές φορές, και αυτό το έχουμε δει και στο παρελθόν, οι συμμαχίες δεν γίνονται μόνο λόγω φιλίας, αλλά και πολλές φορές από φόβο. Βλέπετε λοιπόν πιθανότητα να υπάρξει συμμαχία μεταξύ Κίνας και Ινδίας έτσι ώστε να επικρατήσουν κάποιες θέσεις τους και να εμποδίσουν τις δημοκρατίες του δυτικού κόσμου, τις φιλελεύθερες δημοκρατίες να επιβάλλουν τις θέσεις τους για απελευθέρωση του εμπορίου. Πρόεδρος, από εδώ και πέρα ο χρόνος ομιλίας περιορίζεται σε δύο λεπτά. Από το ΕΛΚ είναι ο επόμενο ομιλητή. Πραγματικά από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ καταρχήν κύριε Επίτροπε για το ξεκίνημα αυτών των διαπραγματεύσεων. Ο διάλογος αυτός σαφώς και θα μας οδηγήσει σε νέες εμπορικές δυνατότητες. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της ε, στρατιωτικής συμμαχίας με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα. Θα έλεγα όμως ότι μέχρι τώρα έχουμε διαπραγματευτεί με χώρες που ήταν ελκυστικοί εταίροι καθότι είχαν μικρότερες αγορές από εμάς, τα συστήματα κανόνων και ρυθμίσεών τους δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένα όσα τα δικά μας. Ήμασταν, αν θέλετε, ο δυνατός εταίρος. Σήμερα όμως αντιμετωπίζουμε έναν πολύ δυνατό εμπορικό εταίρο, μια μεγάλη αγορά, τη δυνατότερη και τη μεγαλύτερη αγορά και για μας το θέμα αυτό είναι θέμα επιβίωσης. Μιλήσαμε για άλλες πτυχές που θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτήν την ε, διαπραγμάτευση με πολλές διαφορετικές ε, συνιστώσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι 27 κράτη, 28 μάλιστα κράτη και αυτό μπορεί σαφώς να μας αποδυναμώσει. Το είδαμε παραδείγματο χάρη αυτό όταν διαπραγματευόμασταν για το θέμα άκτα. Κύριε Πίτροπε, σέβομαι πολύ τις προσπάθειές σας, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τα κακά αποτελέσματα δεν είναι κάτι που σήμερα μπορούμε να το αποκλείσουμε. Το κεφάλαιο που αφορά παραδείγματο χάρη τις επενδύσεις. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι είναι οι στόχοι των Αμερικανών. Είδαμε με την άκτα ότι πολλές από αυτές τις αρχικές τους ε, ε, προθέσεις τις είχαν κρύψει. Πώς λοιπόν εμείς μπορούμε να συγκλίνουμε όταν υπάρχουν τόσο πολλά και διαφορετικά και αντικρώμενα συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Βέρνα από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Καταρχήν και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί ήσασταν σαφέστατος όσον αφορά το περιεχόμενο αυτών των διαπραγματεύσεων Μιλάμε για εμπορικέ αλλαγέ, μιλάμε για επενδύσεις και θα πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι για την ευθύνη που εμείς σαν Κοινοβούλιο και η συγκεκριμένη Επιτροπή πρέπει να αναλάβει. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι παρόμοια με αυτή που έδεκανε η κυρία Σάκε. οι πολιτείες στην Αμερική που όπως ξέρετε πολλές φορές έχουν διαφορετικά πρότυπα, διαφορετικές ρυθμίσεις. Παραδείγματο χάρη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα στην Καλιφόρνια και διαφορετικά στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Την πράξη λοιπόν, τι κάνουμε εμείς, με ποιον διαπραγματευόμαστε, με το ομοσπονδιακό κράτος και πώς αποφεύγουμε συγκρούσεις και εντάσεις. Επίσης, για το Μεξικό έχουμε την παλιά συμφωνία, την οποία θέλουμε να ανανεώσουμε και θα πρέπει εδώ να δούμε ότι όλα εξελίσσονται εκ παραλίλου με την διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένε Πολιτείες, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τη συμφωνία με το Μεξικό. Ευχαριστώ. Thank you. Ο Πολ Θέλω να ρωτήσω ε, τον Επίτροπο. Φαντάζομαι ότι θα έχετε δει από τον Μάρξ Σπόξ από τους Δημοκράτες ε, απευθύνθηκε και στο Κογκρέσο και αναφέρθηκε στα κύρια συμφέροντα ε, των ε, Ηνωμένων Πολιτειών και καταλαβαίνετε ποια είναι τα επιθετικά συμφέροντα των μεγάλων εταιριών των Ηνωμένων Πολιτειών στις διαπραγματεύσεις. Ε, θα αναφερθώ σε τρία πράγματα. Καταρχήν, στο να υπάρχουν μικρότερα εμπόδια για τα αμερικανικά γεωργικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά και ε, επίσης η ίδια διατύπωση χρησιμοποιείται και στην έκθεση της ομάδας, της υψηλής ομάδας εργασίας. Αυτό τι σημαίνει ε, ότι θα υπάρχουν περιορισμοί σε ε, κάποια φάρμακα που χρησιμοποιούνται στα πουλερικά, στο βόλιο κρέας. Ε, τι λέτε ότι όλα αυτά δεν είναι στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ισχυρή προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και λένε ότι είναι το αντιγνωστικό πλεονέκτημα της Αμερικής, η διανοητική διοκτησία και πάλι έχω μια ανησυχία ότι αυτό είναι το μέσο μέσω του οποίου η άκτα ή παρόμοιες διατάξεις μπορούν να μπουν την πίσω πόρτα υπάρχει ένα κενό μεταξύ της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της, ε, τη θέση της πλειοψηφία ε, της κυβέρνησης ε, στη ΣΥΠΑ για το θέμα της προστασίας των δεδομένων και της πνευματικής διοξίας. Το βλέπουμε αυτό στο PNR, στο SWIFT και στην ACTA και πώς θα γίνει σεβαστή η θέση του Κοινοβουλίου και επίσης τονίζουν την ε, ρυθμιστική συμμόρφωση και λένε ότι δεν θα πρέπει να αποδυναμωθούν οι ρυθμιστικές δεσμεύσεις όπως είναι μέσω της υιοθέτηση της αρχής της πρόληψης. Επομένως ε, ε, θα γίνει αυτή η συμμόρφωση προς τα πάνω ή προς τα κάτω και μήπως μέσω αυτής της συμφωνίας που βάζουμε εμείς τα δικά μας πρότυπα. Κύριε Κέλλερ, από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Πριν κάνω τις ερωτήσεις, θέλω να τονίσω ότι οι πράσινοι δεν είναι κατά του εμπορίου καθόλου. Είμαστε υπέρ ε, του δίκαιου του θεμητού εμπορίου και για όλες, ε, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσης, ε, πρέπει να δούμε ποιος επωφελείται και ποιος χάνει από μια εμπορική συμφωνία και πρέπει να ίσως κλείσουμε αυτές τις διαφορές, να τις ισορροπήσουμε. Τώρα, στις ερωτήσεις μου είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό και εκείνη η γνώμη να υποστηρίζει μια τέτοια συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είναι το σώμα που εκλέγεται απευθείας ε, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, εκλέγεται απευθείας από το λαό και η εντολή δίνεται από το Συμβούλιο, προτείνεται από την Κομισιόν. Και ποιο ρόλο λοιπόν σχεδιάζεται να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε την ε, εντολή πριν να λάβει απόφαση το Συμβούλιο. Θα μπορούσαμε να έχουμε και εμεί ένα ψήφισμα, μια γνωμοδότηση που θα ληφθεί υπόψη. Γιατί είμαστε τμήμα της κοινή γνώμης, αλλά και τη διαμορφώνουμε. Και νομίζω ότι αν ε, μας έχετε πει του σκάφους θα είναι σημαντικό. Όπως είπε και ο Πίτερ, θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα διασφαλίσετε ότι μπορούμε να νομοθετήσουμε ε, σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς. Πώς θα διασφαλίσετε ότι μπορούμε να νομοθετήσουμε σε σχέση με τους περιορισμούς, όπως σας είπα, ε, για τα πνευματικά δικαιώματα όταν μιλάμε για τις ανοιχτέ βιβλιοθήκες, ε, γιατί φαίνεται να επιμένουν ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες επ' αυτού. Μπορείτε να επαναλάβετε την τελευταία ερώτηση, δεν κατάλαβα. Πώς θα διασφαλίσετε ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να νομοθετήσουμε για τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις ε, για το copyright για τις βιβλιοθήκες, το χάρη, να μπορούν να υπάρχουν ε, αντίγραφα στις βιβλιοθήκες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε στις διαπραγματεύσεις TPP φαίνεται να έχουν μία τάση να περιορίσουν ακόμη περισσότερο αυτούς τους περιορισμούς. Και τελευταία ερώτηση, μεταρρύθμιση στην προστασία των δεδομένων. Ε, είναι, βλέπετε, ποιες σύγκρουσεις βλέπετε στον τομέα αυτό με τους Αμερικανούς. Πρόεδρος, ε, μάλιστα σημειώσαμε τις δεσμεύσεις των Πρασίνων προς το εμπορίο, αλλά μέχρι τώρα έχετε καταψηφίσει όλες ε, τις εμπορικές συμφωνίες. Η κυρία Σαρνές από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Σημεία, καταρχήν πολιτικό σχόλιο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για να είναι καλή η συμφωνία να εμπλακούμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με ένα ενιαίο μέτωπο. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε πολιτικά ανάντι. Νομίζω ότι το συνειδητοποιείται αυτό. Πρέπει να συνεργαστούν κομισιόν, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μην υπάρχει απόκληση και να έχουμε ένα νέο μέτωπο στις διαπραγματεύσεις απέναντι στον Ομπάμα που θα δεσμεύεται από το Κογκρέσο. Έτσι λοιπόν πρέπει η Ευρώπη να είναι ισχυρή και ενωμένη. Δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τις πολιτισμικές διαφορές. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, όχι μόνο γιατί υπάρχει πίσω από αυτό ένα κοινωνικό μοντέλο και το θέμα της ε, πολιτισμικής διαφοράς, αλλά είναι και το οικονομικό ζήτημα που τίθεται εδώ. Πώς εσείς ε, συλλαμβάνετε το ζήτημα αυτό, πώς μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ. Εμείς έχουμε υπογράψει τη χάρτα της UNESCO, οι ΗΠΑ όχι. Πώς βλέπετε λοιπόν το θέμα της ε, αποδοχής από τους Αμερικανούς αυτής της πολιτισμικής διαφοράς εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να δώσουμε αξία σε αυτή την ποικιλομορφία και όχι να πάμε σε μια μορφή πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης. Τρίτον, πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι το θέμα των προτύπων. Θα έχουμε μια αμοιβαία αναγνώριση ή προσέγγιση των προτύπων αναγκαστικά. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά αυτό το θέμα. Ο κ. Σούλτς μίλησε για απογκασμοποίηση των προτύπων. Καθώς ε, μιλάμε για δύο πολύ σημαντικέ αγορές, μπορεί να φτάσουμε σε αυτό και τότε θα τεθεί το θέμα της ποιότητα και του περιεχομένου των προτύπων. Εσεί πώς το προσεγγίζετε το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω την επόμενη ομιλήτρια. Πίτερ Στάσνε από το ΕΛΚ. Τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν από δύο εβδομάδες ε, παρακολουθούσα πάρα πολύ προσεκτικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον Καναδά που περίμεναν ε, ε, νέα Νομίζω ότι ήσασταν στην Οτάβα και στην Ουάσιγκτον ε, την ίδια εβδομάδα πριν από δύο εβδομάδες. Ελπίζαμε και εμεί να υπήρχαν κάποια ε, τελευταία νέα, κάποια νέα, όπως και στον Καναδά, γιατί είχε υποθεί ότι δεν θα υπάρξει έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης των και Ενωμένων Πολιτειών εκτός, ε, και, εκτός εάν ολοκληρωθεί η ΣΥΤΑ. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο ποια είναι η γενική σας θεώρηση των πραγμάτων και πού πιστεύετε ότι βρισκόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να θέσω ένα ερώτημα στον Επίτροπο. Άλλωστε είμαι και ο εισηγητής για αυτό το θέμα. Κάποιες από τις ερωτήσεις έχουν ήδη τεθεί, οπότε δεν θα επιμείνω. Θα αρκεστώ σε τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, ε, δύο ευρείας πολιτικής σημασίας. Συχνά, ο τύπος παρουσιάζει τους Ευρωπαίους ως το δαίμονα αυτών των διαπραγματεύσεων. Πράγματι ισχύει αυτό και αν όχι, για ποιο λόγο πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι εμείς είμαστε ο δαίμον στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σας. Δεύτερον, δύο επιπλέον μήνες ε, από, από ό,τι προβλεπόταν ε, χρειαστήκαμε για την δημοσίευση της συγκεκριμένης τελικής έκθεσης. Ποιες ήταν οι δυσκολίες, για ποιο λόγο έγινε αυτό. ποιες ήταν οι προϋποθέσεις ε, και από τις δύο πλευρές ε, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα ότι υπάρχει περιθώριο επιτυχούς και φιλόδοξης συμφωνίας ε, όπως αναφέρεται στην τελική αυτή έκθεση. Και τρίτη και τελευταία ερώτηση. Είναι σαφές ότι τα υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά μέτρα ήταν πολύ σημαντικά στο πρώτο αυτό στάδιο και θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά και δύσκολα θέματα των διαπραγματεύσεων. Πώς έχουν προχωρήσει οι δεσμεύσεις, αν έχουν προχωρήσει μεταξύ των δύο πλευρών. Και τώρα, σύμφωνα με την ελληνική έκθεση και τα δύο μέρη συμφωνούν ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και σε διεθνή πρότυπα, όπως επίσης και σε επιστημονική αξιολόγηση κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή πλευρά θα εγκαταλείψει την ε, παραδοσιακή, την παραδοσιακή βασισμένη στην πρόληψη προσέγγιση για να είναι πιο υπέρ τέλος πάντων των Αμερικανών από ό,τι συνήθως ε, ε, ισχύει ε, και από ό,τι συνήθως ακούμε από την ευρωπαϊκή πλευρά για το θέμα αυτό. Και τέλος η τελική έκθεση λέει και παραθέτω ότι εκτός από την συνέχιση της προσπάθειας συμφωνίας θέλουμε να κάνουμε σημαντική πρόοδο και από σχετικά πρώιμο στάδιο ε, σε σχέση με τα υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά μέτρα και σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο και των δύο πλευρών. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό, ποια είναι τα ενδεχόμενα νομοθετικά και διαδικαστικά ζητήματα τα οποία επισήμως δεν αποτελούν τμήμα της συμφωνίας αλλά προκύπτουν και έχουν σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι αυτό το θέμα των φυτοϊγειονομικών και των υγειονομικών μέτρων θα είναι ένα επίμαχο θέμα των μελλοντικών συζητήσεων και πιστεύω ότι πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τι διακυβεύεται εν προκειμένου. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μας. Ε, κύριε Επίτροπε, ξέρω ότι έχετε λίγο χρόνο. Διαλέξτε αν θέλετε, αν δεν μπορείτε να τις απαντήσετε όλες, τις σημαντικότερες ερωτήσεις. Ναι, πρέπει να είμαι λίγο σύντομος γιατί με περιμένει κάποιο στο γραφείο μου. Αλλά θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν ακριβέστερος. Να βρω το χαρτί μου πρώτα. Κύριε Καμάλ, είναι γεγονός ότι δεν του αρέσουν οι γεωγραφικές ενδείξεις των Αμερικανών. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφέ. Έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση για τις μάρκε για τα εμπορικά σήματα. Δεν μας αρέσει πολύ το γεγονός, για παράδειγμα, ότι στη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη είχαμε μια πολύ καλή προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε και με τους Αμερικανούς. Πήρε χρόνια όμως να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να έχουμε τις γεωγραφικές ενδείξεις και δεν, δεν προσπαθώ να κρύψω τη διάσταση απόψεων που υπάρχει από αυτού. Για την άκτα νομίζω ότι έχω ήδη δώσει πολύ σαφή απάντηση. Δεν εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οριοθετήσει Δεν, δεν μπορούμε εμεί να οριοθετήσουμε από ποια στιγμή και μετά ξεπερνάμε το όριο. Κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε για την άκτα, αλλά νομίζω ότι για την ώρα όχι. Απ' την άλλη, οι Αμερικανοί λένε ότι πρέπει να ε, συζητήσουμε και το θέμα των καυσίμων. Τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις πρέπει να γνωρίζουμε ότι παίρνουν συνήθως πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια και ότι έχει νόημα να έχουμε βέβαια μια περιεκτική συμφωνία. Εντάξει, υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές να προχωρήσουμε. Κατά πόσο τώρα το κάνουμε αυτό για να είμαστε φιλικοί ή δίκαιοι, είναι ένας από τους ε, ουσιώδεις ε, ρόλους ε, των κρατών γιατί ε, βέβαια πρόκειται για αποκλειστική αρμοδιότητα ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών της και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αυτή την ευθύνη και εμείς την έχουμε και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά ναι, ως προς τις αξίες οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πολύ πιο κοντά σε εμά από ότι άλλοι, άλλες εμπορικές ε, ομάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε διαφορές. Μαζί τους βέβαια. Κυρία Ζαλεύσκη, μην υποτιμάτε το βαθμό ποικιλότητα στις ίδιες τις Ηνωμένε Πολιτείες. Τεράστιες διαφορές υπάρχουν και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι είναι μικρότερες οι διαφορές αυτές από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν όμως έχει κανείς βλέπει τα πράγματα από μακριά, έχει πάντα την εντύπωση ότι είναι ομοιογενή και όσο πλησιάζει κανείς, τόσο περισσότερες διαφορές ανακαλύπτει. Το ίδιο ισχύει για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Τώρα, κατά πόσο εμείς είμαστε σε πιο αδύναμη θέση, γιατί να είμαστε σε πιο αδύναμη θέση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εντάξει, είναι ε, σκληροί διαπραγματευτές, βέβαια, και εμείς είμαστε όμως, οπότε πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας βοηθήσει σίγουρα. Το ερώτημα τώρα του κυρίου Λάγκε. Αυτά τα πρότυπα για την αυτοκινητοβιομηχανία είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικά αν υπάρχουν διαφορές ε, μεταξύ του κρατικού και του ομοσπονδιακού επίπεδου που δημιουργούν εμπόδια, τότε πρέπει και αυτά να τα ε, εξετάσουμε. Όπως για παράδειγμα πρέπει να κάνουμε με τις δημόσιες συμβάσεις. Και σίγουρα είναι ένας ε, παράγοντας που περιπλέκει τα πράγματα. Μεξικό. Υπάρχει σχέση και δεν υπάρχει παράλληλα. Έχουμε μία συμφωνία με το Μεξικό. Μεξικανοί μας ε, ζήτησαν να την ε, επικαιροποιήσουμε τη συμφωνία και είπαμε ότι Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Επίσης μας ζήτησαν από την αρχή να είναι τμήμα των διαπραγματεύσεων για το TPIP και εγώ είπα ότι δεν νομίζω ότι αυτό είναι ρεαλιστικό. Δεν θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο. Απλούστατα. Είναι όμως μια περιεκτική η συμφωνία με τι Ηνωμένες Πολιτείες που θα είχε αντίκτυπο στο Μεξικό λόγω των συνδέσμων ε, με το Μεξικό και για τον Καναδά ισχύει αυτό, αλλά δεν χρειάζεται να τα αιμαδοποιούμε όλα αυτά μαζί ε, γιατί δεν θα υπάρχει η δυνατότητα διαχείριση του πλέον. Τα, βλέπω λοιπόν αυτά ω αλληλουχία, ε, βλέπω ότι υπάρχει ένα αντίκτυπο και για την ε, αυτοκίνητο βιομηχανία και το λέω αυτό παράδειγμα. Κύριε Μέρφυ, αν αποκλείεται η Γεωργία, Δυστυχώς δεν ήσασταν παρόν ε, στην πρώτη ε, στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Είπα όμω ότι είναι σημαντικό τμήμα των διαπραγματεύσεων και για την άκτα ε, εξέφρασα σαφέστατα τις απόψει μου. Κατά πόσο εκτό μικροφώνου ο κύριο Μέρφυ τη συμπληρωματική ερώτηση που δεν ακούμε. Η απάντηση είναι ναι, γνωρίζω αυτή την επιστολή. Την επιστολή που αναφέρατε Και σωστά αναφέρεται αυτό το ε, αριθμητικό στοχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τον φυσβητώ αυτό. Όμως, οι διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή έχουμε μία εντολή. Είναι διαπραγμάτευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Αμερικανικής Κυβέρνησης. Πολλές απόψεις θα ακουστούν. Βεβαίως θα τι ε, λάβουμε υπόψη, θα τις σημειώσουμε και θα εξασφαλίσω ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα έρχομαι και σε επαφή με το Κογκρέσο. Έχω σκοπό να πάω εκεί, να ε, συζητήσω και με μέλη του Κογκρέσου και με γερουσιαστές. Ε, δεν χρειάζεται να με πείσετε λοιπόν γι' αυτό. Ξέρω λοιπόν την επιστολή και ξέρω τι ζητούν. Είναι επιθετικά συμβαίροντα αυτά και εμείς θα κάνουμε το ίδιο. δεν υποβαθμίζουμε το επίπεδο προστασίας. Το ότι εναρμονίζουμε δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζουμε, αλλά από την άλλη... Να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα με τις νόρμες και με τα πρότυπα. Αυτή τη στιγμή τα αποκτά κανείς και μπαίνει στη διαδικασία, είναι πεπισμένος ότι τα δικά του είναι τα καλύτερα. Βέβαια, η άλλη μέρα έχει την ίδια άποψη για κάτι που είναι διαφορετικό. Οπότε Γι' αυτό πιστεύω ότι για τα ρυθμιστικά πρότυπα θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος. Και αν θέλουμε πραγματικά κάτι επαναστατικό, πρέπει στο μέλλον να στοχεύουμε σε κοινέ διαδικασίε για την αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει κανεί κάτι, γίνεται θρησκεία. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συζητήσει κανεί το θέμα τη θρησκεία. Κυρία Κέλλερ, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την εντολή. Όταν στέλνουμε εντολή στο, στο Συμβούλιο, θα στείλουμε και στο Κοινοβούλιο. Είμαι διατεθειμένος να τη συζητήσω μαζί σας και ε, βεβαίως έχετε την ελευθερία και περιμένω να το κάνετε, να ε, ε, ψηφίσετε ένα ψήφισμα για αυτό το θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το συζητήσω διεξοδικά, αλλά στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματο. Και το χρονοδιάγραμμα νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σαφές. Σα το κατέστησα σαφέ. Μπορούμε βέβαια να το κάνουμε αυτό που θέλετε εντό του χρονοδιαγράμματο. Κανένα πρόβλημα. Θα έχετε τη δυνατότητα να το συζητήσετε. Θα το έχετε στη διάθεσή σα. Και βεβαίω μπορείτε να υποβάλλετε και ψήφισμα. Φορέ το είπα. Ποια είναι η άποψή μου για την άκτα. Και δεν θα το ξαναπώ. Ούτε έχω σκοπό να ξαναμπεί η άκτα από την πίσω πόρτα στι διαπραγματεύσει. Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, ξέρετε ότι υπάρχει μια συνεχή συζήτηση για, τα ε, ε, για το θέμα αυτό στι ΗΠΑ. Μία συζήτηση τώρα για αυτό το θέμα και δεν νομίζω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή ο, ο σωστός τρόπος θα ήταν να το ε, θέσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι μία άλλη πορεία αυτή και Θα συνεργαστώ πολύ στενά με την ε, Επίτροπο Ρέντινγκ που είναι και υπεύθυνη για το θέμα αυτό. Ελπίζω πριν από το τέλος των διαπραγματεύσεων να καταλήξουμε σε μια κοινή κατανόηση. Αυτό άλλο θέμα βέβαια. Όμως δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα πάντα γιατί ήδη έχουμε αρκετά να εξετάσουμε. Αναφερθήκατε στις εξαιρέσεις Εγώ δεν διάβασα αυτό το κομμάτι της, ε, του TPP. Δεν μπορώ να σας δώσω λοιπόν μια συγκεκριμένη απάντηση. Η πηγή έμπνευση είναι παρόμοια και θα δούμε μετά πώ ακριβώ θα το διαπραγματευτούμε με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά ευχαρίστω να επανέλθω στι λεπτομέρειε ε, γραπτώ σε σχέση με αυτά που ρωτήσατε. Κυρία Ντεσαρνέε. Βεβαίω είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ενιαία θέση και να έχουμε και την υποστήριξη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο ε, δεν είναι φτιαγμένο για να έχει ενιαία θέση. Πρέπει να αντικατοπτρίζει τις διάφορες απόψεις και μετά θα δούμε πού είναι η πλειοψηφία. Ελπίζω ότι η πλειοψηφία θα είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω τουλάχιστον ελπίδες. Πολλέ ελπίδε. Δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε την πολιτική μας για την πολιτιστική ποικιλομορφία. Ξέρω είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, παρά το γεγονό ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πολύ το φοβόμαστε. Εντάξει, άλλο θέμα αυτό, δεν βλέπω για ποιο λόγο μια παγκοσμιοποίηση πολιτιστική θα είχε ως αποτέλεσμα μια αμερικανική ηγεμονία. Εγώ βρίσκω ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός θα τα πάει τόσο άσχημα. Έχουμε τόσα πολλά πλεονεκτήματα. Αλλά τέλος πάντων η ιδέα μας δεν είναι να αλλάξουμε την πολιτική ως προς την πολιτιστική ποικιλομορφία. Κύριε Στάζνη, για τον Καναδά. Είναι απλή η απάντηση. Πήγαμε, Πήγαμε πρώτα στη Ουάσιγκτον, μετά πήγαμε στην Οτάβα. Αυτά που ήταν στο διαπραγματευτικό τραπέζι εμένα δεν μου άρεσαν και γι' αυτό ακριβώς δεν συμφώνησα. Ήταν απλό και του στόπα. Πρέπει να λάβουν επιπρόσθετα μέτρα, να κάνουν επιπρόσθετα βήματα και αν δεν τα κάνουν δεν θα υπάρχει συμφωνία. Γιατί νομίζω ότι η συμφωνία θα έπρεπε να υπάρχει μόνο όταν είναι καλή. Και για πολλά ζητήματα πρέπει να κάνουν και άλλα βήματα. Βέβαια θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μαζί τους και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις σύντομα, αλλά η άποψή μου είναι ότι μια συμφωνία πρέπει να είναι καλή. Μόνο όταν είναι καλή η συμφωνία, τότε τη συνάπτουμε. Και αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή δεν προμηνύουν καλή συμφωνία. ο μόνος, η μόνη σχέση μεταξύ τους, ε, μεταξύ Ουάσιγκτον και ε, Οτάβα, ε, και Οτάβας είναι ότι είναι κοντά. Ότι το πιο, ο πιο εύκολος τρόπος να πάει κανείς στην Οτάβα είναι να περάσει από τη Ουάσιγκτον και το ανάποδο. Τέλο πάντων, είναι κοντά, καμιά ώρα τέλο πάντων και ε, αυτό είναι ο μόνο στόχο. Αυτό είναι το μόνο κοινό στοιχείο. Τα σχόλια είναι εκτό μικροφώνου του κυρίου Στάσνη. Η απάντηση πάντως είναι δεν γνωρίζω τη δήλωση αυτή και θα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση ε, αν έγινε τέτοιου δήλωση ενδεχομένως να υπήρξε παρε... παρεξήγηση. Προσπαθούμε να έχουμε μια συμφωνία με τον Καναδά και μια συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες σχέσεις για συγκεκριμένα θέματα ως προς την αυτοκινητοβιομηχανία για παράδειγμα, ε, γιατί ο Καναδάς σημαίνει το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, αλλά εκτός από αυτό δεν υπάρχουν άλλα κοινά στοιχεία. Κατά πόσο ε, ζητάει ε, πράγματα, ζητούν πράγματα οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, Προφανώ. Διαφορετικά δεν θα είχαμε διαπραγματεύσει. Για ποιο λόγο διαφορετικά να μπούμε σε διαπραγματεύσει, αν δεν υπάρχουν αιτήματα. Κάποιοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είπαν σαφέστατα ότι πιστεύουν ότι είναι πολύ σημαντικό. Ε, ναι, αλλά αν ο κύριο Ομπάμα, που είναι ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ενδιαφερόταν για μια συμφωνία μαζί μα, δεν νομίζω ότι θα άρχιζε τι διαπραγματεύσει. Για ποιο λόγο πήρε επιπλέον δύο μήνες. Ε, είναι απλή η, η απάντηση. Ε, υπήρχε μια μεταβατική περίοδος μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Αυτός νομίζω ότι είναι ο πραγματικός λόγος. Τώρα, η παραδοσιακή, αν θέλετε, ορολογία των συμφωνιών ε, του ΠΟΕ και αν θα την ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ναι, αυτή θα ξαναχρησιμοποιήσουμε και για αυτήν την συμφωνία. Έχουμε λοιπόν συνεχίσει την επεξεργασία των επιπλέον αυτών θεμάτων και όπως είπατε και εσείς Πρόκειται καθαρά για δυσκολίες και για τομείς για τους οποίους θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Το θέμα, αν θέλετε, του πώς μπορούμε να αποφύγουμε να επεκταθούν όλες αυτές ε, οι περιπτώσεις στην εσωτερική αγορά. Είδατε τι έγινε με το κρέας ε, των αλόγων, παραδείγματο χάρη. Και εκεί υπάρχει θέμα. Αλλά και για την ε, σπογκώδη εγκεφαλοπάθεια, παραδείγματο χάρη, θα υπάρξουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις τους επόμενους μήνες. Δεν είναι η τελευταία συζήτηση που έχουμε για το θέμα αυτό, ελπίζω. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όποιες και να είναι οι θέσεις ε, των μεν και των δε. Και υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Θα πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα ουσιαστικά θέματα, στα αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά. Και για μένα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε αυτές τις δύο αγορές, να δείξουμε ότι με, μόνο με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνουμε την θέση μας παγκοσμίω. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές, αλλά παρόλα αυτά είμαστε οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες και κοινωνίες με ελευθερία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν τεχνικά, υπάρχουν πολιτιστικά προβλήματα, διαφορές νοοτροπίας, αλλά σε επικεντρωθούμε στα κοινά μας όποια και να είναι η πολιτική μας, φιλοσοφική μας άποψη και από όποια χώρα και αν προερχόμαστε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Είναι όντως η πρώτη συζήτηση, θα ακολουθήσουν πολλές για τη συμφωνία αυτή και σας εύχομαι επιτυχία και επιτυχή συμφωνία. Θα παρακολουθήσουμε και θα στηρίξουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις παρόλο που ίσως δεν θα είμαστε παρόντες στην ε, σύναψη της συμφωνίας. Very good. Ladies and gentlemen, there is. Yes. There is still much work to do. Έχουμε ακόμα πολλά θέματα για σήμερα το πρωί. Καθίστε παρακαλώ. Those who are leaving the room, do it. Βγείτε γρήγορα από την αίθουσα με ησυχία. Only a small remark to... Και θα ήθελα να αντιδράσω σε κάτι που είπε πολύ σωστά ο Επίτροπος ότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά 200% τις επενδύσεις και τα εμπορικά θέματα, τις εμπορικές συναλλαγές. Είναι λοιπόν κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα και άλλες επιτροπές, τη γεωργία, τις μεταφορές, ΣΥΜΚΟ. Εμείς από την αρχή σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να συνεργαστούμε με τις άλλες επιτροπές, γι' αυτό και εγώ έγραψα στους προέδρους των άλλων αρμόδιων επιτροπών. Από την αρχή ήδη συνεισφέρουμε όλοι την επόμενη εβδομάδα. Εγώ θα τους ε, γράψω πάλι και θα οργανώσω μία μόνιμη, αν θέλετε, συνεργασία με τους σκιώδες ηγητές, με μένα, για το θέμα αυτό. Έτσι ώστε να μπορέσουν όλες οι υπόλοιπες επιτροπές να συνεισφέρουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην επεξεργασία αυτού του θέματος. Και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Καθώς είμαι σίγουρος ότι εμείς θα παίξουμε διευθυντικό, ηγετικό ρόλο. Ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν στο θέμα 16 που είναι το πλαίσιο για τη διαχείριση της ε, δημοσιονομικής ε, ευθύνης. Πρόκειται για ένα σχέδιο έκθεσης. Ε, ήδη έχει γίνει η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριος Ζαλεύσκη είναι ο εισηγητής μας και έχετε την έκθεση αυτή στους φακέλους σας. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και βεβαίω θα ακούσουμε τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς μετά από τα εισαγωγικά μου σχάλια θα αναγκαστώ να φύγω. Και δεν το κάνω επειδή δεν σέβομαι τα μέλη της Επιτροπής, αλλά γιατί κανονικά έπρεπε να είχαμε αρχίσει πριν από μία ώρα. Και εγώ με περιμένει ένα αεροπλάνο και πρέπει να φύγω, να γυρίσω στην Πολωνία. Δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει ο Πρόεδρος. Ζητώ λοιπόν συγγνώμη, αλλά ξέρω ότι όλες οι προτάσεις σας και όλες οι απαντήσεις σας και τα σχόλιά σας θα μου μεταφερθούν με ακρίβεια. Έχουν υποβληθεί τροπολογίες όσον αφορά την πρόταση Επιτροπής για τη θέσπιση πλαισίου διαχείρισης οικονομικής ευθύνης σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών. Οι πολιτικές ομάδες έχουν συνεισφέρει με προτάσεις και γνωρίζετε όλοι το σχέδιο έκθεσής μου, διότι έχει διανεμηθεί στους κοιόδες εισηγητές και ακολούθησαν συζητήσεις της ε, προηγούμενης εβδομάδας. Και Ήδη έχω κάνει κάποιες σημαντικές ε, αλλαγές. Όπως σας είπα, κατά τη διάρκεια την πρώτη μας συζήτηση, πιστεύω πραγματικά ότι το κείμενο της Επιτροπής είναι καλά διαρθρωμένο, ισορροπημένο κείμενο, γι' αυτό και υιοθέτησα μια προσέγγιση που βασίζεται μάλλον στην τροπολογία, τροποποίηση του κειμένου και όχι σε καμιά ριζοσπαστική αλλαγή. Γι' αυτό και έχω υποβάλει αυτές τις αλλαγές. Δεν θα υποβληθεί μεγάλος αριθμός τροπολογιών, αλλά θα περιοριστούμε σε αυτές τις ε, αλλαγές που είναι πολύ συχνά γλωσσικές, ε, θέματα διαφήνειας, σαφήνειας, συγγνώμη, διαφάνειας του κειμένου. Το άρθρο 8, παραδείγματος χάρη, και η παράγραφος 2 χρήζουν ε, κάποιων τροποποίησεων. Αποφάσισα λοιπόν να αλλάξω τη διατύπωση, να γίνει πιο συγκεκριμένη, γιατί πιστεύω ότι η αρχική διατύπωση δεν είναι καθόλου σαφής και στο σημείο C και στο σημείο D. Σκοπός μου είναι ξεκινώ από μία ασάφεια όσον αφορά τις διάφορες προτάσεις εδώ που μπορούν να ερμηνευθούν με πολλούς τρόπους και να ξεκαθαρίσω λίγο τους όρους και τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό και αναφέρομαι εδώ στις ε, διάφορες ε, παρατηρήσεις που είτε έχουν γίνει είτε μπορεί να προκύψουν. Μπορεί να προκύψουν λοιπόν διάφορες ε, περιπτώσεις διαφορών, των οποίων η επίλυση μπορεί να επηρεάσει την μελλοντική ερμηνεία το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 9 παράγραφος 2. Πιστεύω ότι η αρμοδιότητα της Επιτροπής εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί. Αναφερόμενοι εδώ στις διάφορες διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. Και οι δύο αυτές παράγραφες θα πρέπει σαφώς να διατυπωθούν με πιο συγκεκριμένο τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών. Άρθρο 18. Διαιτητικό κόστος. Κόστος της ε, διαδικασίας. Και εδώ υπάρχει μια σάφια στην ερμηνεία. Εκφράσαμε επίσης και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη δική μας δράση καθώς και όλη την απαραίτητη πληροφόρηση που χρειάζεται για όλες αυτές τις διαιτητικές διαδικασίες που τυχόν θα προκύψουν. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Μπορείτε να μας εγκαταλείψετε για να μην χάσετε το αεροπλάνο σας. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ τον εισηγητή, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή που μας ε, ενημερώνει όσον αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε αυτό το θέμα. Η ομάδα των σοσιαλιστών παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον και θα στηρίξουμε μάλλον το κείμενο αυτό. Δεν έχουμε ακόμα φτάσει στην τελική μας θέση βεβαίως. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι στο σχέδιο αυτό κανονισμού που κοιτάμε τις ε, υποχρεώσεις, ε, τις οικονομικές υποχρεώσεις Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις των σοσιαλιστών όσον αφορά την επίλυση αυτών των διαφορών και τους μηχανισμούς επίλυσης. Κάτι που κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να το δούμε ξεχωριστά στην συζήτηση αυτού του κανονισμού. Ανησυχούμε, παραδείγματο χάρη, εδώ βεβαίως μας έχει δώσει κάποιες εγγύσεις η Επιτροπή, αλλά Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να δούμε το θέμα της αρμοδιότητας του κοινοτικού νομοθέτη όσον αφορά θέματα παραδείγματος χάρη ε, δημόσιου συμφέροντος και εδώ αναφερόμαστε παραδείγματος χάρη σε θέματα καπνού, τσιγάρων για επιχειρήσεις τρίτων χωρών και ξέρουμε ότι σε τέτοιες διαιτητικές ε, διαδικασίες θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη διατύπωση έτσι ώστε να καλύψουμε όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν. Επίσης ανησυχούμε, τουλάχιστον όταν διαβάζω το κείμενο, γιατί μπορεί αυτός ο μηχανισμός να δημιουργήσει δικαιώματα σε κάποιες ε, επιχειρήσεις τρίτων χωρών όσον αφορά τις επενδύσεις. Εδώ βεβαίως δεν μπορούμε να επικαλεστούμε τις ε, διατάξεις ISDS, αλλά θα πρέπει αυτό να ξεκαθαριστεί από την Επιτροπή. Γιατί οι οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το ISDS δεν θα πρέπει εδώ να παραμείνουν ασαφείς, ιδιαίτερα όταν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε διαιτητικά δικαστήρια. Ξέρετε ότι οι δυνατότητες αυτές μπορούν να δώσουν σε αλλοδαπούς επενδυτές περισσότερα δικαιώματα από αυτά που έχουν οι εγχώροι επενδυτές, οι επενδυτές ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή Απλώς αναφέρω τα προβλήματα και είναι πιο εύκολο να αναφέρει κανείς τις τυχόν δυσκολίες παρά να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Αλλά πραγματικά εδώ θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να μην υπάρχει μεταξύ των επενδυτών από τρίτες χώρες, τους ξένους δηλαδή επενδυτές, ε, σε σχέση με τους ε, χώριους. Ο εισηγητής κάλυψε κάποια θέματα. Εμείς όμως οι σοσιαλιστές θέλουμε να αναφέρουμε πρώτον τη διαφάνεια, δηλαδή η διαδικασία να είναι όσο διαφανής γίνεται, θα κάνω μια γραπτή πρόταση με περισσότερες λεπτομέρειες και δεύτερον ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο για όλες αυτές τις υποθέσεις και το ίδιο πρέπει να ισχύει για τα κράτη-μέλη και για το Συμβούλιο. Εξίσου θα πρέπει να ενημερώνεται και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ λοιπόν την Επιτροπή για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και βεβαίως ε, και τον εισηγητή, ο οποίος λείπει, αλλά είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Κάζακ από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ. Λείπει η σκιώδη συγγητριά μας. Θα παρουσιάσω όμως ε, εγώ την άποψή της. συντομία, ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για το εξωτερικό του έργο για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Πρόκειται για το δεύτερο νομοθετικό φάκελο για την πολιτική προστασία ε, των επενδυτών ε, που μας απασχολεί σε αυτήν την Επιτροπή Διαπραγματεύσεις ε, με την Κομισιόν και το Συμβούλιο για τον κανονισμό grandfathering των κεκτημένων δικαιωμάτων. Δεν ήταν εύκολε. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή που απευθύνθηκε στην κρατή μέλη σε έγκαιρο στάδιο για να ακούσει τα σχόλιά τους. Παρ' όλα αυτά, Ω Κοινοβούλιο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η αρμοδιότητα σε αυτό το τομέα πολιτικής έχει μετακινηθεί στην Ένωση με σαφήνεια και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σεβαστούν τη Λισαβόνα. Η αρχή τη ενότητα στην εξωτερική εκπροσώπηση ε, καλύπτει και τις επενδυτικέ πολιτικές και η Κομισιόν πρέπει να υπερασπιστεί αυτή την αρχή. Η Γενική Αρχή για αυτή την ε, πρόταση είναι σαφής και σωστή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει όταν ε, μιλάμε για δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κράτος μέλος πληρώνει όταν ε, θίγεται. Το κράτος μέλος όμως πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Αυτός ο αυτό το νομοθέτημα θα πρέπει να φέρει ασφαλή δικαίου για την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη όταν δεν είναι προφανέ σε ποιον αναλογεί ευθύνη εκ πρώτη όψεων. Στην ε, πρότασή τη όμω η Κομισιόν μπορεί να πηγαίνει κάπω πολύ μακριά στην ε, προσπάθεια να αναλάβει ευθύνη όταν δεν είναι ξεκάθαρη η ευθύνη που αναλύει ευθύνη. Έχοντα κατά νου τον κοινωνισμό περικεκτημένων δικαιωμάτων, θα πρέπει να βρούμε μια καλή ισορροπία με το με των κρατών μελών να υπερασπίσουν τον εαυτό του όταν οι πράξει του όταν οδηγούνται στο δικαστήριο για τις πράξεις τους. Ε, ε, εμείς θεωρούμε ότι η κατεύθυνση του εισηγητή είναι σωστή σε κρίσιμα άρθρα όπως το άρθρο 8 ή το άρθρο 9 που αφορά τις διαδικασίες βρίσκει ο εισηγητής καλύτερη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων κρατών ομελών και της Κομισιόν ενώ επιβεβαιώνει τις γενικές αρχές που υπάρχουν στην πρόταση της Κομισιόν. Επίσης, το άρθρο 18 για την ε, καταβολή του κόστους ε, της επίλυσης διαφορών είναι καλύτερη πρόταση του εισηγητή από τις Κομισιόν. Σε αυτό το σχέδιο έκθεσης, επίσης, θα πρέπει να δούμε και άλλα άρθρα, όπως είναι το άρθρο 3 το άρθρο 11 και κάποια ακόμη. Αν υπομονούμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή για τις τροπολογίες ε, και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κάζακ. Η κυρία Κέλλερ από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ζαλεύσκη, κυρίως επειδή συνεργάστηκε με τους σκιώδεις σε πρώιμο στάδιο. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία μας. Εξέπληξε όταν ε, εξετάσαμε την έκθεση μας εξέπληξαν κάποιες αντιφάσεις που φαίνεται να υπάρχουν ε, με το grandfathering, ε, τα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά και τη θέση του κυρίου Ζαλευσκή για το grandfathering. Γιατί ε, εκεί ήθελε να υπερασπίσει τις διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνα, που είναι σήμερα φυσικά Δίκαιο Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταφέρει την αρμοδιότητα από τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω στην έκθεση βλέπουμε ότι ορισμένα αυτά, από αυτά είναι αντιφατικά. Έτσι λοιπόν να ξαναδούμε το άρθρο 8 και τι τροπολογίε 2 και 5 που πιστεύω ότι δεν προσδιορίζουν ακριβώς ε, τα πράγματα αλλά μεταφέρουν την αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη σε τομείς που δεν συμφωνούμε. Προτείνει ο εισηγητής να υπάρχει μία απόφαση στην περίπτωση του ενάγοντα, σε περίπτωση που έχει χαθεί υπόθεση άρθρο 2, άρθρο 8 παράγραφος 2, ενώ η Κομισιόν σωστά προτείνει ότι θα πρέπει να δράσει η Ένωση αν πρόκειται να παρουσιαστούν παρόμοιες αξιώσεις υπό την ίδια συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι είναι μόνο αναδρομική η υπεράσπιση της έντοσης. Αν ε, είχαμε υπεράσπιση από τα ίδια τα κράτη-μέλη, θα είχαμε διαφορετικό επίπεδο υπεράσπισης σε παρόμοιες υποθέσεις. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Και είναι σημαντική αυτή η διαφορά γιατί είναι πιθανό να προκύψουν τι καταστάσεις στα σε κράτη-μέλη ε, όπου υπάρχει προσφυγή κατά αυτών για τον τρόπο που έχουν εφαρμόσει την νομοθεσία. Και σε ό,τι αφορά την τροπολογία 19 για τις υποχρώσεις υποβολής εκθέσεων, δεν ε, ξέρω αν θα πρέπει να ζητήσουμε μια πρώτη μόνο μετά από πέντε έτη. Δηλαδή θα έχει περάσει και μία ολοκληρή θητεία, ενώ η Κομισιόν προτείνει τρία έτη για την περίοδο αυτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιλέξουμε την πιο σύντομη χρονική περίοδο και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα τρία έτη στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο αργότερα. Επίσης, θέλω να επανέλθω και στο γενικό πρόβλημα που έθεσε ο Ντεβιτ Μάρτιν, που έχουμε η πράσινη με τον κανονισμό αυτό και δεν λύνεται από την Επιτροπή ούτε από τον εισηγητή. Το συζητήσαμε και στις συναντήσεις των σχεδόν εισηγητών ότι η πρόταση υποθέτει ότι υπάρχει οικονομική ευθύνη της Ένωσης, ακόμη και αν η εξίωση καταφέρεται κατά της νομοθεσίας της Ένωσης, ε, που φυσικά έχει ελεγχθεί προσεκτικά από εμά και από άλλους, για να μην είναι ασύμβατη με το διεθνές διεθνό δίκαιο. Και επίσης η εφαρμογή τη παρακολουθείται προσεκτικά. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να συμφωνήσουμε με μια τέτοια προπόθεση με τέτοια υπόθεση καταρχήν ε, θα οι τροπολογίες μας θα ακολουθήσουν την ιδέα ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφανθεί επί αυτού του θέματος και οι μελλοντικέ επενδυτικές συμφωνίες δεν θα πρέπει να προβλέπουν οποιαδήποτε οικονομική ευθύνη της Ένωσης ενώ της Ένωσης επενδυτή που πηγαίνει πέρα των εφιστάμενων μηχανισμών στη συνθήκη και αντιστεί στην ομολογία του δικαστηρίου. Δεν υπάρχει λόγος οι επενδυτέ από τις τρίτες χώρε να δικαιούνται να διτούν ε, διεθνεί διαιτητέ ε, και να θεωρούν υπεύθυνη την Ένωση για νομοθεσία που έχει υιοθετηθεί από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ δεν αναγνωρίζουμε τέτοιο δικαίωμα στους Ευρωπαίους επενδυτές, δύναμη δηλαδή του Ευρωπαϊκού Δικαίου να ζητήσουν αντιστάθμιση δηλαδή το ελάχιστο που, χρησιμο... που απαιτείται για τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας ε, ε, κατά επιπόλαιων αξιώσεων ε, βλέπουμε να υπάρχει ε, τέτοιες Βλέπουμε να υπάρχουν τέτοιε περιπτώσει σε τρίτες ε, χώρε σε περίπτωση νομοθεσία στον τομέα τη υγεία, παραδείγματο χάρη περιβολητικής νομοθεσία. Και δεν πρέπει ε, τέτοια νομοθεσία να παρεμποδίζεται από κάποιε επιπόλε αξιώσει. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο θέμα αυτό και επίση δεν πιστεύουμε ότι είναι της μηχανισμό φιλτραρίσματο, δηλαδή να βάζουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκεί ανάμεσα θα ήταν ε, κάτι απαράδεκτο για του εταίρου γιατί η έρωση και τα κράτη-μέλη χαίρονται υψηλότερο επίπεδο της ε, δέουσας επιμέλειας στις δικαστικές διαδικασίες και παραμένει πάντα η δυνατότητα οι επενδυτές από τρίτες χώρες να προσφύγουν και στα εθνικά δικαστήρια. Και έχω την εντύπωση από προηγούμενες συζητήσεις ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι συμφωνούν με αυτή την ανησυχία, συμμερίζονται αυτή την ανησυχία. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δράσουμε έχοντας αυτά κατά νου σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτς από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομολογώ ότι η ομάδα μου έχει κάποια προβλήματα με, αυτόν, με αυτή την πρόταση κανονισμού, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εξή ζήτημα. Για ποιο λόγο πρέπει να εισαγάγουμε, εκτός από το ε, δικαστικό σύστημα να υπάρχει ένα επιπλέον ε, συμβούλιο όπως ε, αυτά τα πάνελ επίλυσης διαφορών. Είμαι πεπισμένος ε, ότι σε, όλε, σε όλα τα νομικά συστήματα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο δικαστικής δικαιοσύνης και δεν ισχύει νομίζω μόνο για τις χώρες του ΩΣΑ αλλά και για άλλες χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να επανεπισημάνω Μία θέση που έχει πολλές φορές ε, ακουστεί της πλειοψηφίας ε, του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου ότι το δικαστήριο θα έπρεπε να είναι υπεύθυνο για ζητήματα επίλυσης τέτοιου είδους διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών και όχι τα ειδικά αυτά πάνελ. Πρέπει να δούμε δηλαδή τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα ε, όταν ένα κράτος θέλει να ε, καταγγείλει ε, μία επένδυση σε κάποιο, σε κάποιο από αυτά τα πάνελ επίλυσης διαφορών. Πρέπει να το δούμε αυτό. τα πάνελ επίλυσης διαφορών επενδυτών κρατών δεν ικανοποιούν κανένα, καμία από τις προϋποθέσεις. Ε, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας, κάτι το οποίο ε, ανέφεραν και, άλλες, ε, και άλλοι συνάδελφοι. Η έλλειψη κατάρτισης για αποφάσεις που υπερβαίνουν τα καθαρά επιχειρηματικά συμφέροντα. Και υπάρχει επίσης και το, ε, η, μη δυνατότητα υποβολής ε, έφεσης. Οπότε με απασχολεί πραγματικά η εισαγωγή αυτών των πάνελ, αυτού του μηχανισμού, ε, ως αντικατάσταση της νομικής διαδικασίας της συνήθους που έχουν στη διάθεσή τους οι κυβερνήσεις και όπως αναφέρεται στο σχέδιο γνωμοδότησης, στο σχέδιο έκθεσης του ε, συναδέλφου, για τον οποίο τον ευχαριστώ βέβαια, γιατί έχει προσπαθήσει να λάβει υπόψη πολλά πολλά στοιχεία, πολλές απόψεις. Δεν υπάρχει όμως αυτό το ερώτημα των συνεπειών της προτινόμενης νομοθεσίας σε σχέση μεταξύ, ε, της, σχέσης, μεταξύ της σχέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη-μέλη. Βλέποντα λοιπόν την περίπλοκη πραγματικότητα, λαμβάνοντα υπόψη την περίπλοκη πραγματικότητα τη μεταγραφή ε, μια Ευρωπαϊκή οδηγία στα κράτη-μέλη, ε, υπάρχουν ορισμένα εκκρινή ζητήματα σε σχέση με την νομοθεσία, παρά το γεγονό ότι υπάρχει μια προσπάθεια από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα αμβλύνει τα προβλήματα αυτά. Υπάρχει το θέμα λοιπόν ε, της, του, του κατά πόσο ε, η Επιτροπή ε, ή το κράτος πρέπει να αναλάβει ε, δράση ή αν υπάρχει μία απόφαση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το πάνελ πρέπει, όταν, όταν πρέπει το πάνελ ας πούμε να, να αποζημιώσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ε, ποιος θα τα πληρώσει αυτά, αυτός ο προϋπολογισμός από πού θα βγει. Ε, η ομάδα μου λοιπόν έχει πάρα πολλές απορίες για, τις οδηγίες αυτές, για την οδηγία αυτή. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Dartmouth. Συγγνώμη κύριε Φιέλ, είναι προηγούμενο, νομίζω. Εγώ πάντοτε υποχωρώ μπροστά στον κύριο Φιέλνερ, αλλά τώρα δεν θα το κάνω. Όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό προκύπτει από τη συνθήκη της Λισαβόνας και είδα την αιτιολογική έκθεση με ιδιαίτερη προσοχή και είδα μια πρόταση που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης να συμπεριλαμβάνει τις συμφωνίες για όλα τα θέματα σε σχέση με τις ξένες επενδύσεις και τις ξένες άμεσες επενδύσει. Ε, δείχνει η τερά, την τεράστια αλλαγή που εισήγαγε βόνας. Αυτό σημαίνει και θυμάμαι τα σχόλια του ε, Jim Murphy που ήταν ε, ε, ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Ζητημάτων της κυβέρνησης των εργατικών το γνωρίζει αυτό ο κύριος Μάρτιν, ε, είχε πει ότι είναι ένα εγχείρημα εκαθάρισης. Ε, νομίζω ότι οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος θα έλεγε ότι ε, ελπίζω ότι ο κύριος Μάρτιν είναι σε αυτή την κατηγορία των λογικών ανθρώπων, θα έλεγαν ότι είναι μια τεράστια παρεξήγηση, μια κακή ερμηνεία προς τους Βρετανούς. Να μπω τώρα σε πολλές λεπτομέρειες. Ε, λέει στην αιτιολογική έκθεση ότι η πρόταση δεν έχει υποβληθεί σε ε, αξιολόγηση αντικτύπου και γιατί όχι. Θα έπρεπε να είχε γίνει κάτι τέτοιο γιατί είναι πραγματικά μια σημαντική νομοθεσία και δεν έχει γίνει καμία τέτοιου είδους μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου. Επίσης λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πολλές συναντήσεις με εκπροσώπους των κρατών μελών στις προετοιμασίες ε, της πρότασης και ότι οι απόψεις λήφθησαν δεόντως υπόψη στη συνημένη πρόταση. Ακόμη και με τα στάνταρ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, είναι πολύ αόριστα όλα αυτά. Και θα ήθελα να μου πείτε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό αυτές τις συναντήσεις που έλαβαν ε, χώρα με τους εκπροσώπους των κρατών μελών και κατά πόσο όντως ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις τους. Τώρα, όταν πρωτοβλέπει κανείς αυτή την πρόταση, είναι ένα παράδειγμα που μας θυμίζει πολλά ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συγκεκριμένη Επιτροπή. Είναι μια συνεχής επίθεση, μια συνεχής υποβάθμιση, αποδυνάμωση ε, της ακαιρεότητας του κράτους έθνους, ε, κάτι με το οποίο εγώ διαφωνώ απολύτως. Μάλιστα. Κοιτάξτε, η Επιτροπή μας ε, δεν είναι ένα βήμα για βρετανοβρετανικές ε, μάχες. Ε, τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Φιέλνερ. Κοιτάξτε, δεν θέλω να με, να με ξεχάσουν. Αυτό ήταν το μόνο πράγμα. Δεν θα ήθελα να με ξεχάσετε, γι' αυτό διαμαρτυρήθηκα. Δύο πράγματα θα ήθελα να θέσω. Η κυρία Κέλλερ και ο κύριος Μάρτιν τα είπαν και μου έκανε λίγο εντύπωση. Μου θύμισε Κάτι διαφορετικό. Η κυρία Κέλλερ είπε ότι βλέπουμε κατά πόσο η νομοθεσία που προτείνουμε συμπορεύεται με τις ε, συνέπειες ε, στο εμπόριο κλπ. Ε, το... Τα νέα προϊόντα καπνού, για παράδειγμα, είναι ένα, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης. Προσπαθήσαμε να το δούμε αυτό σε σχέση με την οδηγία ε, για τα προϊόντα καπνού και αυτό θα ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα για το κατά πόσο ε, θα έπρεπε ε, να ελέγχεται η προτινόμενη νομοθεσία με υπάρχουσε εθνικέ νομοθεσίε. Γιατί μπορεί να υπάρξουν όλο και περισσότερο τέτοιου είδου εμπορικέ διαμάχε και συγκρούσει. Και εμεί είμαστε, υποτίθεται, οι ειδικοί για αυτά τα θέματα. Ίσως οι συντονιστέ θα έπρεπε να προβληματιστούν από αυτού κατά πόσο θα έπρεπε εμείς να συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση λίγο παραπάνω. Πρόεδρος, κύριε Φιέλνερ, πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Νομίζω ότι και άλλε επιτροπές θα έπρεπε να σκέφτονται τι εμπορικέ συνέπειες ζητημάτων που ε, συζητούν στις ε, επιτροπέ του. Να ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εδώ ο συνήθις εκπρόσωπος. Ξέχασα κάποιον. Α, ξέχασα κάποιον που ήταν και πρώτος στη λίστα μου. Τον κύριο Λάγκε, συγγνώμη σας ξέχασα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι, όπως ξέρετε οι τελευταίοι έσονται πρώτοι όπως λέει και η Παλαιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη, συγγνώμη. Θα ήθελα να σας πω καταρχήν ότι η σχέση μεταξύ των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε σχέση με τις αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τι καλύπτεται και τι δεν καλύπτεται από την κοινοτική νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παραδείγματος χάρη το θέμα ενός ε, πανεπιστημίου που ε, βρίσκεται σε μια διαμάχη με το κράτος το οποίο βρίσκεται. Εκεί δεν υπάρχει αρμοδιότητα κοινοτική ή παραδείγματο χάρη στη Γερμανία αποφασίσαμε όλες οι, πυρηνικές, οι μονάδες πυρηνικής ενέργειας να ε, παύσουν τη λειτουργία τους. Και εδώ μπορεί να υπάρξει προσφυγή παραδείγματο χάρη των επενδυτών. Και εδώ, και εδώ, βάσει της συνθήκης, δεν υπάρχει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν υπάρχουν τα προβλήματα και εδώ θα πρέπει να επεξεργαστούμε το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ, Επιτροπή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Θα σε ευχαριστούμε που μας καλέσατε με σκοπό να σχολιάσουμε το σχέδιο κειμένου, να απαντήσουμε. Καταρχήν να η συνεργασία μας με τον εισηγητή, με την Επιτροπή, με το Κοινοβούλιο για την περαιτέρω επεξεργασία του κειμένου ε, ήταν πολύ καλή. Κοιτάξαμε πολύ προσεκτικά την πρόταση κανονισμού, αλλά και γενικότερα το θέμα της ε, επίλυσης διαφορών, το κατά πόσο τα εργαλεία που διαθέτουμε είναι επαρκή γενικότερα για να καλυφθούν ε, θέματα που μπορεί να προκύψουν και να οδηγήσουν σε διαφορές. Πριν πω όμως ε, συγκεκριμένα στο σχέδιο κειμένου και στον κανονισμό. Σας παρακαλώ πολύ να είστε σύντομοι, λέει ο Πρόεδρος. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Όσον αφορά τώρα την επίλυση διαφορών που έχουν σχέση με τους επενδυτές, θα ήθελα να σας πω καταρχήν ότι υπάρχουν οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως οι δικαιωτικές ε, αρχές καλύπτουν τις περισσότερες από αυτές ε, τις ε, διαφορές. Εδώ βλέπουμε δηλαδή το θέμα των επενδύσεων και των επενδυτών. Έχουμε τα εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ε, Ευρωπαίων επενδυτών. Υπάρχουν όμως παρόλα αυτά περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να λυθούν διακρατικά. Γι' αυτό και χρειάζεται να υπάρχει και αυτή η επιπλέον ε, δυνατότητα επίλυσης των διαφορών. Τώρα, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, βεβαίως είναι το ε, κατεξοχήν δικαιοδοτικό όργανο όπως ξέρετε, οι συμφωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε φορά επιλύονται αλλού εκτός Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εδώ θα πρέπει να δούμε για αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και τμήματα αυτών των διεθνών συμφωνιών κάθε φορά ορίζεται το αρμόδιο δικαιωτικό όργανο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να εξετάσουμε αυτές τις περιπτώσεις και να δούμε πώς μπορεί αυτή η ουσιαστική προστασία την οποία αναφέρουμε σε όλες μας τις συμφωνίες να εμπεριέχεται στη διατύπωση η ισορροπία των, της προστασίας των δικαιωμάτων μεταξύ των επενδυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει εδώ να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν αρκετές ε, διατάξεις που να αναφέρουν αυτήν ακριβώς εδώ την πτυχή της προστασίας. Δεύτερον, τι έχουμε να πούμε όσον αφορά τη διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αναφέρατε αυτό, γι' αυτό και εμείς ε, ε, διαπραγματευόμαστε στα πλαίσια των ε, Ηνωμένων Εθνών, διεθνείς διαδικασίες ε, διαφάνειας για τις εμπορικές συναλλαγές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και αυτή εδώ η συμφωνία να περιέχει κάποιες διατάξεις που αφορούν τη διαφάνεια. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επικαλυστούμε στη συμφωνία για να αυξηθεί η διαφάνεια, μηχανισμοί διαιτητικής επίλυσης των διαφορών, πρόκειται και για κάποιες επιπλέον ε, δυνατότητες, μια πολύ σημαντική προσθήκη, ένα νέο στοιχείο σε αυτή τη συμφωνία. Το θέμα τώρα των ε, άλλων ε, δικαστηρίων, αν η προσφυγή γίνεται ελεύθερα ή αν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ε, πιστεύω ότι εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα επιμείνουμε σε αυτό να υπάρχουν δεσμευτικές ε, διατάξεις για το θέμα της επιλογής των ε, διαδικασιών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δημόσιο συμφέρον, παραδείγματο χάρη. Επαναλαμβάνω, εδώ θα πρέπει οι διατάξεις να είναι δεσμευτικές. Όσον αφορά τις τροπολογίες που πρότεινε ο εισηγητής και τα σχόλια που ακούστηκαν για τον κανονισμό. Καταρχήν, ευχαριστούμε τον εισηγητή, καθότι συμφώνησε με την γενική δομή της πρότασης της ε, ε, Επιτροπής. Αυτό μας ε, οδηγεί σε εξοικονόμηση χρόνου έγιναν συναντήσεις ε, με τους εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου εκ των προτέρων και νομίζω ότι αυτή η καλή προετοιμασία μας οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Έγιναν ε, συναντήσεις τεχνικών εμπειρογνωμόνων στη φάση της ε, σύνταξης αυτού του κειμένου και πραγματικά η διαδικασία η προετοιμασίας ήταν πολύ σημαντικό, ήταν πολύ προσεκτική και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι οι τροποποιήσεις θα είναι περιορισμένες. Θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας με τον εισηγητή, με τους κοιόδες για όλα τα σχόλια που κάνατε σήμερα. Ανεπίσημα, αλλά και εδώ στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Τώρα, όσον αφορά το σχέδιο των την τροπολογία 5. Εδώ έχουμε παρουσιάσει ένα νέο κείμενο με περισσότερες κατηγορίες αξιώσεων. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα σχόλια που κάνατε και νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε τη διατύπωση για να δούμε ότι καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις τις οποίες σκεφτόμαστε. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες αξιώσεων. Ίσως εδώ το κείμενο πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο όσον αφορά παραδείγματος χάρη τις ε, διαβουλεύσεις που θα πρέπει να γίνονται ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πολλές παράλληλες διαδικασίες για παρόμοιες υποθέσεις. Τώρα, τα θέματα που θίξατε όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των επενδυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ δεν υπάρχει συγκεκριμένη διατύπωση, αλλά μπορούμε εδώ να καθοδηγήσουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα κράτος μέλος, αλλά επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι των κρατών μελών. Εδώ λοιπόν όταν αναφερόμαστε στο, ε, τα, στα υπέρμετρα συμφέροντα, το υπέρμετρο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέψτε μου να πω ότι θα πρέπει να είναι και προς συμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην περιορίσει την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 14 και 15 άλλες δύο τροπολογίες εμείς ε, στηρίζουμε αυτές τις επιπλέον προτάσεις, δηλαδή να μπορεί να ζητηθεί περισσότερη ενημέρωση για μια υπόθεση, περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία και επαναλαμβάνω προσβλέπουμε σε περισσότερη διαφάνεια σε δημόσια έγγραφα, δημόσια στοιχεία, δημοσίευση των ε, στοιχείων και να παραμένουν ε, απόρριτα μόνο τα καθαρά εμπιστευτικά στοιχεία και έγγραφα και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ε, Επιτροπή ε, την δική σας για την περαιτέρω πρόοδο των ενεξελίξη υποθέσεων και διαφορών. Όσον αφορά λοιπόν τις απαιτήσεις για περισσότερη διαφάνεια, με μεγάλη χαρά θα κοιτάξουμε τις προτάσεις σας. Νομίζω ότι απάντησα σε όλα τα σχόλια. Άκουσα και σχόλια για το 8 και το 9, τα δύο άρθρα. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε μια πιο ισορροπημένη διατύπωση όσον αφορά την συνοχή στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου έτσι ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους στις ε, εκρεμείς διαδικασίες. Επαναλαμβάνω ότι όταν πρόκειται για θέματα εθνικά, όπως αυτά που αναφέρατε, της πυρηνικής ενέργειας ή ενός πανεπιστημίου στο εσωτερικό ενός κράτους, ναι, Εάν ένας επενδυτής θεωρήσει ότι το κράτος μέλος συμπεριφέρεται α, παραβιάζοντας μία συμφωνία, εδώ απλώς για να απαντήσω στην παρατήρηση που κάνατε, σε αυτή την περίπτωση, όταν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός, μπορεί ο εν λόγω επενδυτής να επικαλεστεί ότι το κράτος μέλος δεν λειτουργεί μόνο σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση δηλαδή να εξεταστεί αν πρόκειται καθαρά για θέμα εθνικής νομοθεσίας ή αν παραβιάζεται η κοινοτική νομοθεσία και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ξεκαθαρίσουμε όταν πρόκειται για περιπτώσεις επενδύσεων που εμπίπτουν στην κοινοτική νομοθεσία, στην κοινοτική αρμοδιότητα, δηλαδή κάτι που απαιτεί ενότητα και εξωτερική εκπροσώπηση. Σε άλλες περιπτώσεις, οι διαφορές μπορεί να επιληθούν σε εθνικό επίπεδο, από τα εθνικά δικαστήρια. Και αυτό βεβαίως και όσον αφορά τις ε, οικονομικές επιπτώσεις μια τέτοιας διαδικασίας η οποία αναλαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο. Ο κανονισμός, εν πάση περιπτώσει, Εάν προκύψουν τέτοιες διαφορές μεταξύ επενδυτών και εθνικών αρχών, μπορεί να καλύπτονται από την κοινοτική αρμοδιότητα. Το θέμα είναι ότι οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν τις πτυχές τις οποίες αναφέρεται αυτή η διαφορά. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε εάν ε, όπως έγινε στην περίπτωση της Σιγκαπούρης, ε, του Καναδά, αν στην ε, εμβέλεια της συμφωνίας εμπεριέχονται και αυτές οι διαφορές. Και αυτό είναι θέμα αξιολόγησης. Αυτά κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις. Με μεγάλη χαρά θα επεξεργαστούμε περισσότερο τις προτάσεις αυτού του κειμένου και θα επανέλθουμε εδώ όταν μας καλέσετε. Σας ευχαριστώ. Ο εισηγητής είπαμε έφυγε. Δεν μπορεί λοιπόν να απαντήσει στις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής. Αλλά βεβαίως θα επανέλθουμε στη συζήτηση αυτού του θέματος όταν συζητήσουμε τις τροπολογίες. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 26 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο το 17 και το 18. Um, since we'll not have the time to deal... Καθώς δεν θα έχουμε το χρόνο να δούμε σήμερα όλα τα σημεία στην ημερήσια διάταξη, ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε μόνο αυτό. Και να αφήσουμε τα επόμενα για να τα συζητήσουμε σε επόμενες συνεδρίες. Λοιπόν, σημεία 17 και 18 πρόκειται για την αποκατάσταση της πρόσβασης της ΜΜΑΡ στις γενικευμένες δεσμολογικές προτιμήσεις. Ο κύριος Ντεβιτ Μάρτιν είναι ο εισηγητής. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα θυμούνται οι συνάδελφοι σε προηγούμενη συζήτηση ότι το Διεθνέ Γραφείο Εργασία και του UC μα είχαν ε, αναφέρει ότι υπήρχαν εξελίξει στη Βερμανία για την εξάλληψη τη ε, καταναγκαστική εργασία. Ε, δεν ισχυριζόμαστε βέβαια ότι έχει εξαλειφθεί εντελώ, αλλά βάσει των συζητήσεων αυτών και ευρύτερων διαβουλεύσεων. Έχω καταρτήσει το σχέδιο έκθεση μου σε μια πρόταση τη Κομισιόν και προετοίμασα και, μια, ένα συνοδευτικό ψήφισμα. Καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στην Βερμανία έχουν γίνει πραγματικά βήματα για τον εκδημοκρατισμό και την επίλυση των συγκρούσεων. Όμω εξακολουθεί να ε, υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει στη χώρα. Η απόσυρση της χώρας από την πρόσβαση στο σύστημα γεννητημένων προτιμήσεων έγινε είναι βάσει κάποιων κριτηρίων του ΔΟΕ. Η Κομισιόν προτείνει την αποκατάσταση της πρόσβασης της Βρυμανίας στο γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων ε, καθώς η καταναγκαστική εργασία δεν αποτελεί πλέον σοβαρή και συστημα... δεν συμβαίνει πλέον σοβαρά και συστηματικά. Συστήνω λοιπόν στο σχέδιο εκθεσίσμου μου να επικυρώσουμε την πρόταση της Κομισιόν γιατί πρόκειται για ένα απλό φάκελο. Δεν προτείνω κάποιε τροπολογίε για την πρόταση της Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά δεν πιστεύω ότι από το μηδέν μπορούμε να πάμε ε, στο τέλειο εν μία νυχτή. Έτσι λοιπόν θα πρότεινα να υπάρχει και ένα συνοδευτικό ψήφισμα στην έγκρισή μας που θα θέτει κάποιες προϋποθέσεις. Υπήρξε σαν κυρώσει που έχουν επιβληθεί από το 1996 από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Βερμανία και αν ε, λάβουμε υπόψη την ευάλωτη κατάσταση στην οποία είναι η χώρα σήμερα, κατανοούμε ότι πρόκειται για μια μοναδική περίπτωση. Επομένω, καλωσορίζω τη δήλωση τη ε, κυρία Άστον ότι θα υπάρξει μια task force τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα για την ενδυνάμωση τη οικονομική συνεργασία. Ε, τώρα, ε, πρέπει να δούμε ε, ότι ε, έχουμε δει επενδύσεις από βιομηχανίες, από κλάδους στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και από άλλες χώρες, τη Βερμανία, οι Ηνωμένε Πολιτείες, οι Άπωνες και άλλοι όλοι προσπαθούν να μπουν στην αγορά της Γερμανίας. Ε, καθώς υπάρχει έλλειψη στη χώρα, ε, δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα του συνέρχεστε και του συνεταιρίζεστε ε, και υπάρχει και πρόβλημα με τις εξωτερικές βιομηχανίες, πρέπει να κινηθούν πολύ προσεκτικά οι ευρωπαϊκοί επενδυτές, όμως έχουμε ε, τις ε, αρχές, ε, τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς υπάρχουν και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει εμείς να προωθήσουμε τις βελτιστές πρακτικές στην Βερμανία. Στο σχέδιο ψηφίσματος προτείνω να υπάρξει ένας μηχανισμός προκειμένου να μπορούν να κάνουν δηλώσεις ε, και να καταγγέλουν ε, οι επιχειρήσεις ε, το τι συμβαίνει στην Βερμανία. Έχουμε το ίδιο σύστημα για τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Στέλνουν τις κατευθύνσεις τους γραμμές στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ. μπορούμε να θεσπίσουμε ότι θα συλλέγονται οι εκθέσεις συλλογικά, πόσες πληροφορίες θα συλλέγονται και αν θα είναι υποχρεωτική, υποχρεωτικός ο χαρακτήρας. Η Βερμανία ε, βρίσκεται σε μια κατάσταση μεταρρυθμίσεων. Έτσι λοιπόν πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόζονται οι βέλτιστες κριτικές. Ε, θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με τη Βερμανία και θέματα διαφάνειας. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι οδηγίες καλύπτουν μόνο ορισμένου εξορεκτικούς τομείς και δεν απαιτούν αποκαλύψεις για πληρωμές που καταβάλλονται στις κυβερνήσεις. Για να κλείσω, Πρόεδρε, καλωσορίζω την πρόταση της Κομισιόν να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο σύστημα προτιμήσεων, γιατί είναι ένα λογικό βήμα κατόπιν της άρσης των κυρώσεων της ΔΟΕ, αλλά νομίζω ότι πρόκειται και για ένα λογικό βήμα στη Βερμανία για τη μείωση της φτώχειας και την οικονομική μεγέθυνση και ελπίζουμε έτσι να υποστηρίξουμε και την μετάβαση προς τη δημοκρατία. Βέβαια, η Βερμανία είναι σε πολύ ευάλωτη την κατάσταση και εξακολουθούν να υπάρχουν εκεί παραβιάσεις των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει, ε, να θεσπίσει ένα πλαίσιο για εταιρική κοινωνική ευθύνη, έτσι ώστε και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν ε, σε ένα θετικό περιβάλλον. Μάλιστα, ευχαριστούμε από το ΕΛΚΟ, κ. Φιέλνερ. Ευχαριστώ. Καταρχήν για την απόφαση που πρόκειται να λάβουμε, συμφωνούμε. Δεν έχουμε να συζητήσουμε πολλά επ' αυτού. Νομίζω ότι το έχουμε επιλύσει αυτό με τις προηγούμενες συζητήσεις, όμως μπορούμε να συζητήσουμε τη διατύπωση του ψηφίσματος. Γενικά δεν διαφωνώ επί συγκεκριμένων ε, ζητημάτων, όμως μπορεί να υπάρξουν κάποιες αποχρώσεις. Ακόμη και αν κάποιος διαφωνεί με το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου, εγώ αν ε, το διατύπωνα ο ίδιος το κείμενο θα είχε διαφορετική ισορροπία. Στην παράγραφη 3 έως 10 αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πολύ σημαντική είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά αν δούμε τη Βερμανία, εγώ θα είχα επικεντρωθεί περισσότερο και μπορεί να επανέλθω με τροπολογίες στις μεταρρυθμίσεις ε, στις οποίες έχουν προβεί οι Βερμανοί και τι περιμένουμε, ότι περιμένουμε να παραμείνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις Β. Τι θέλουμε περισσότερο και τι περιμένουμε από αυτούς να πράξουν ε, για να βελτιώσουν την κατάσταση. Έχετε αρκετά στα εκτιμώντας, όμως νομίζω ότι στο διδακτικό του κειμένου θα έπρεπε να επικεντρωθούμε περισσότερο στα θέματα αυτά και μιλάτε για τις ευάλωτες μεταρρυθμίσεις ε, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό το να συνοδεύει αυτή την αποφασία από τη έρετε και κοινωνική ευθύνη. Συμφωνώ μεν, αλλά αυτό δεν ε, είναι σχετικό μόνο με τη Βερμανία. Δεν ισχύει μόνο για τη Βερμανία. Θα έλεγα ότι περισσότερες ε, χώρες CBA, όλα πλήν των όπλων, εντάσσονται σε αυτό. Και έρχομαι στο σημείο 7 γι' αυτό τον ειδικό κεντρικό μηχανισμό. Αφενός, συμφωνώ και το κατανοώ γιατί το προτείνεται. Γιατί η Βερμανία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και δεν μπορεί κάποιος ε, εν μία νυχτή να περάσει από τη χειρότερη κατάσταση στην καλύτερη. Όμως, ε, εδώ δεν μιλάμε για τη Βερμανία, αλλά για τις εταιρείε και για το τι θα πρέπει να κάνουν επομένως. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα απομόνωνα τη Βερμανία έτσι για το τι πρέπει να κάνουν οι εταιρείε μας. Αν πρέπει να κάνουν κάτι τέτοιο, πρέπει να το κάνουν και τις υπόλοιπε χώρες, η BA που είναι στο καθεστώς, οτιδήποτε πλήν όπλων. Αλλά και ειδικά στην Βερμανία χρειαζόμαστε αυτό το μηχανισμό. Επιφυλάσσομαι λοιπόν να ξανασκεφτώ το σημείο 7 και να επανέλθω, αλλά θα ήθελα να υπάρχει μια ισορροπία σε σχέση με το θέμα των μεταρρυθμίσεων στη Βερμανία. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε σοβαρή πίεση χρόνου. Για να δούμε ποιος είναι ο κατάλογος των ομιλητών. Τρία λεπτά για την κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Σκεφτήκαμε σοβαρά το θέμα αυτό και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υποστηρίζουμε και τη θετική προσέγγιση του κυρίου Μάρτιν. Ακολουθούμε λοιπόν την πρότασή σας ε, για την αποκατάσταση της πρόσβασης, αλλά συμφωνούμε και με τις ανησυχίες σας. Και θέλουμε να υπάρχει αυτό το ψήφισμα και υποστηρίζουμε το περιεχόμενό του αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής Ο κύριος Μόρφη. Ευχαριστώ πολύ. Θα διαφωνήσω. Θα είμαι αυτός που θα διαφωνήσει. Ευχαριστούμε για την έκθεση. Ναι, συμφωνώ ότι έχουν γίνει βελτιώσεις, ειδικότερα στον τομέα της καταναγκαστικής εργασίας, αλλά πρέπει να δούμε τι μήνυμα ε, αποστέλουμε ε, στις πολυεθνικές και σε χώρες που προσπαθούν ε, να πάνε στην ε, Μιανμάρ για πρώτες ύλες. Τι ακριβώς μήνυμα δίνουμε με αυτήν την βιασύνη να επανεισαγάγουμε το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Ναι, υπήρχαν βελτιώσεις, υπήρξαν βελτιώσεις στην καταναγκαστική εργασία δεν ξέρω κατά πόσο είναι αναπότρεπτες αυτές οι πρόοδοι βέβαια, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν για τις εθνοτικές μειονότητες πολλά διαφωνώ με την επανεισαγωγή των προτιμήσεων για την ώρα. Όσον αφορά τώρα το θέμα της καταναγκαστικής εργασίας, νομίζω ότι υπάρχει επαρκής, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ε, συνεχιζόμενης καταναγκαστικής εργασίας για να δικαιολογήσουν τη μη επανεισαγωγή. Ειδικότερα συμβαίνει για παράδειγμα στις ε, στρατιωτικές δυνάμεις και γύρω από αυτές. Πριν από ένα μήνα η ΔΟΕ ε, βοήθησε διαπραγμάτευση ανήλικων ε, τη διαπραγμάτευση για ε, απομάκρυνση ανήλικων ε, ε, στρατιωτικών στις στρατιωτικές δυνάμεις και στην διαδικασία εξόριξης χρησιμοποιούνταν επίσης ανήλικοι, κάτι το οποίο πραγματικά βρίσκω πολύ σημαντικό. Ε, νομίζω λοιπόν ότι το γεγονός ότι υπάρχει κάποια πρόοδος χρησιμοποιείται ως πίεση για άλλα πράγματα. Εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι, υπάρχει καταστολή και νομίζω ότι την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει ε, για τον, ε, ε, του εκτοπισμού 34.000 ατόμων. Νομίζω ότι υπάρχουμε, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη κλιμάκωση όσον αφορά τις εθνοτικές μειονότητες 90.000 άτομα ε, ε, εθνοτικών μειονοτήτων στη, ε, στο βόρειο Μιανμάρ εξακολουθούν να εκτοπίζονται. Νομίζω λοιπόν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και γι' αυτό δεν συμφωνώ με το μεγαλύτερο τμήμα του σχεδίου ψηφίσματος νομίζω ότι θα έπρεπε να πιώσουμε ε, προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που λέει ο κύριος Φιέλνερ, περισσότερες δηλαδή υποχρεώσεις ε, ε, για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την παρουσία τους ε, ε, στο Μιανμάρ. Το δικαίωμα, για παράδειγμα, της απεργίας ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται σεβαστό στην πραγματικότητα και όχι μόνο στη θεωρία. Ευχαριστώ πολύ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία, ο κύριος Κανιάδο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να πω ότι επικροτούμε το, το σχέδιο έκθεσης, το οποίο ε, βέβαια ε, αφορά ε, τη συμμόρφωση με το δίκαιό μας, όπως επίσης και τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. με το σχέδιο ψηφίσματος δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα, το λάβαμε την περασμένη εβδομάδα, θα θέλω όμως να πω ορισμένα προκαταρτικά πράγματα που μπορεί να σας είναι χρήσιμα. Οι συζητήσεις αυτές δεν θα γίνουν στο κενό, αλλά εν ώψη πολλών πρωτοβουλειών της Επιτροπής, όπως η δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον τομέα του αερίου και του πετρελαίου, δύο, παρακολούθηση δεσμεύσεων ε, εφαρμογής των συγκεκριμένων ε, της ε, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, επίσης αποκάλυψη ορισμένων στοιχείων από την κυβέρνηση, όχι μόνο στην εξορεκτική βιομηχανία, αλλά και σε άλλους κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περίπτωση του Μιανμάρ και επίσης επερχόμενη νομοθεσία όσον αφορά τη βελτίωση της διαφάνειας για, για την υποβολή περιβαλλοντικών και κοινωνικών εκθέσεων. Κάτι επίσης πολύ ε, σημαντικό σε σχέση με το Μιανμάρ. Ε, επίσης, η κυβέρνηση του Μιανμάρ είπε προσφάτως στην αρχή του χρόνου ότι σκοπό έχει να ε, προσχωρήσει στην ε, πρωτοβουλία της διαφάνειας για την εξωτερική βιομηχανία. Έχουμε κάποιες ε, πρωτοβουλίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί και κάποιες από τις πρωτοβουλίες αυτές ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν κάποιες από τις ανησυχίες της επαρκώς, ώστε να μην χρειάζεται να ιδρύσουμε άλλους μηχανισμούς που μάλλον δεν θα βοηθήσουν πολύ τους ε, στόχους που θέλετε να επιτύχετε. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί πολλές φορές το λέω. Συγγνώμη, ισχύει, λέει ο Πρόεδρος, ε, το χρονικό όριο και για σας. Μήπως μπορείτε να, να ολοκληρώσετε. Ναι, βεβαίως, θα ήταν χρήσιμο να παραμείνουμε στις συστάσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε ε, σε σχέση με, το με την ομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις. Μιλάω για την, για την αιτιολογική σκέψη 9 και 10. Καταλαβαίνουμε διαφορετικά την, το περιεχόμενο και τη φύση της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ ε, και θα έρθουμε σε επαφή με τον εισηγητή για να το αποσαφηνίσουμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. David, καταληκτικά σχόλια. Ναι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Καταρχά, ε, να ευχαριστήσω την κυρία Κέλλερ για την υποστήριξη. Συμφωνώ ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με ε, το Μιανμάρ, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την εθνική, εθνοτική βία. Το, κατά το θέμα μας είναι κατά πόσο όμως πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΔΟΕ για την άρση των κυρώσεων. Γιατί και εκείνοι μας το συνέστησαν αυτό. Όσον αφορά τώρα το ψήφισμα, επιχειρεί να επικεντρωθεί περισσότερο, Κρίστοφερ, στις ευρωπαϊκές εταιρείες από τη... του Μιανμάρ. αν επανεισαγάγει την εργασία ε, το Μιανμάρ, ε, βεβαίως ε, θα απομακρυνθούν και πάλι, θα καταργηθούν και πάλι οι προτιμήσεις για τη χώρα αυτή. Αυτό που εμείς πρέπει να πούμε νομίζω είναι οι υποχρεώσεις των ευρωπαϊκών εταιριών επειδή ξέρω το περιβάλλον στο οποίο θα πάνε, πρόκειται για μια δημοκρατία ακόμα δύναμη και υπάρχει λίγη παρακολούθηση, νομίζω ότι οι ειδικέ υποχρεώσει σε σχέση με ε, τι ευρωπαϊκέ χώρε, ε, με τι ευρωπαϊκέ εταιρείε, θα πρέπει να υπάρχουν για το Μιανμάρ συγκεκριμένα. Όσον αφορά τώρα την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις σχετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Καλά είναι όλα αυτά. Επίσης το θέμα αυτό δεν είναι... Αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ακριβώς ίδια με αυτά που κάνει ο ΟΗΕ. Από ό,τι κατάλαβα εξακολουθούν να υπάρχουν διαπραγματεύσεις και το θέμα της ετήσιας υποβολής εκθέσεων δεν θα αρχίσει, από... δεν θα αρχίσει παρά μόνο τον Απρίλιο. Είπα όμως ότι οι συστάσεις μας ε, δεν είναι ίδιες με αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με το τι κάνει ο ΙΕ ε, και αναφέρομαι σε σχέση με τις ε, διατάξεις για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πολύ ειδικέ δραστηριότητε στο Μιανμάρ για να εξασφαλίσουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι στο περιβάλλον αυτό και το λέω αυτό σε σχέση με αυτά που είπε και ο Κρίστοφερ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη γνώμη μου είναι μοναδική περίπτωση ε, το Μιανμάρ. Πρόεδρος, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες, στι 6 το απόγευμα. Δηλαδή σε 5 μέρες από σήμερα. Και για το ψήφισμα ισχύουν αυτές ε, οι προθεσμίες. Τα 20 και 21 θα τα αφήσουμε για επόμενη συνεδρίαση. Τότε να πάμε στο 22. Γιάννη Ξαντού. Που είναι ο εισηγητής μας. για την πρώτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις δραστηριότητες των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών. Είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και δίνω το λόγο στον ε, εισηγητή για να μας παρουσιάσει τις απόψεις του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε πολύ μικρό χρόνο, πολύ λίγο χρόνο, αλλά είναι καλό να ξεκινήσει η διαδικασία. Πράγματι βρισκόμαστε σε μια περίεργη κατάσταση γιατί λάβαμε το έγγραφο εργασία της Κομισιόν που παραπέμπει σε αυτή την υποχρέωση με τα κρατή-μέλη να πούνε ουσιαστικά να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ε, θα τους εφαρμογεί τα απαιτούμενα τη συνθήκη σε θέματα περιβάλλοντος, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφάνειας ε, των λογαριασμών τους και είχαμε το πρώτο εγχείρημα. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν το μέσα, μέσα Δεκέμβρη σας έστειλε μια έκθεση, αλλά ήταν προσωρινή προσωρινή έκθεση βάσει του εξή. Δεν μπορούμε ακόμη να αξιολογήσουμε το σύνολο, της κομισι... το σύνολο του έργου τη Κομισιόν για να δούμε τι εφαρμόζουν, αν εφαρμόζουν του ορθού κανόνε ε, στον ΟΣΑ τα κρατημέλη. Έτσι λοιπόν πρέπει να το δούμε αυτό με την γραμματεία τη ΣΥΝΤΑ και δεν ε, κατανοήσαμε ακριβώ το καθεστώ του εγγράφου τη Κομισιόν. Περιμένουμε απαντήσει από την Κομισιόν. Όμω, σήμερα υπάρχουν χώρε που καταβάλουν την προσπάθεια για να προσπαθήσουν ε, να αποδώσουν καλύτερα τον ε, αντίκτυπο των ε, προγραμμάτων των εξαγωγικών πιστώσεων. Βέβαια αυτό είναι ανεπαρκές γιατί στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και αυτό είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα να παρουσιάσουν τις μη χρηματοοικονομικές πτυχές της δουλειάς τους και συγκεκριμένα στα περιβαλλοντικά. Προτείνουμε λοιπόν να έχουμε αυτή τη μήνυα ακρόαση το Μάρτιο που θα μας επιτρέψει μαζί με τους προσκεκλημένους μας ε, είτε από τη ΓΑΜΑ Μάρκετ, από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ θα έχουμε για κάποιον από τον ΩΣΑ και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις ε, μη οικονομικές δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη βάση σας προτείνω να καταρτήσω την έκθεση πρωτοβουλίας και καθώς πρέπει να είμαι πολύ γρήγορα, θα δώσω και τις εμβιώσεις μου σε όλους τους κοιοδησίτες για να καταλάβουν σε ποια ακριβώς κατάσταση βρίσκεται το φάκελος αυτό. Ο πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Έχουμε ένα μισή λεπτό για τους επόμενους ομιλητές. Ξεκινάμε από τον κύριο Μέρφυ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και του Γερμανείς για τον πλέον χρόνο. Πολύ σύντομα, νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε δει σε σχέση με τις εκθέσεις αυτές από τα κράτη-μέλη ότι είναι ανεπαρκής πολύ συχνά έχουμε μεταφορικό εγχείρημα να κάνουμε κλικ, ότι σέβονται τα διάφορα πρότυπα και τους κανόνες. Πολλές ε, εκθέσεις χωρών είναι παρόμοιες. Τους χάρη, ρωτά εδώ στην έκθεση εφαρμόζεται τις κοινέ προσεγγίσεις του ΣΑΣ ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά και την κοινωνική ιδέως επιμέλεια. Ναι, εφαρμόζεται το ένα το άλλο, ναι, ναι πολύ ωραία, τότε τα εφαρμόζουν όλα και είμαστε ικανοποιημένοι. Είναι αναπαρκές. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα αν πρέπει να έχουμε μια πραγματική εποπτεία του τι συμβαίνει. Και κάτι ακόμη σε σχέση με τη χρήση των κοινών προσεγγίσεων του ΩΣΑ. Δεν είναι νέο το έγγραφο, ούτε όλα τα μέλη είναι μέλη του ΩΣΑ όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του ΩΣΑ. Έτσι λοιπόν μήπως θα έπρεπε η Κομισιόν να καταρτήσει ένα έγγραφο ευρωπαϊκό και να χρησιμοποιούμε αυτό αντί της, των κοινών προσεγγίσεων του ΩΣΑ. Τις δέχομαι εγώ τις κοινέ προσεγγίσεις του ΩΣΑ, αλλά θεωρώ ότι δεν επαρκούν. Και εγώ είμαι πεπισμένος, λέει ο Πρόεδρος, ότι σε ένα μισή λεπτό μπορείτε να πείτε αυτά που συνήθως λέτε σε πέντε λεπτά. Ο κύριος να Ευχαριστώ. Καταρχήν, η πρόταση αυτή μας ανησυχεί πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα που έχουμε ξανακούσει. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε γιατί τα κράτη πρέπει να υποχρεούνται να αναφέρουν στην Κομισιόν ε, σχετικά με τις εξαγωγές τους πιστώσεις, αλλά υπάρχει κάτι πιο ανησυχητικό εδώ, Δηλαδή, βλέπουμε εδώ, περιγράψτε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε τη Wills Royce, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο μηχανών jet ε, και τείνουν να χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από εξαγωγικές πιστώσεις. Και εγώ καταλαβαίνω ότι οι πράσινοι που ε, είναι πολύ καλή πολιτική όπως το είναι, όταν οι πράσινοι βάλουν κάτι μέσα που θα καταστήσουν τις εξαγωγές της ε, Βρετανίας σχεδόν αδύνατες. Έτσι λοιπόν, ε, ε, εγώ βλέπω κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνει ούτε τώρα, ούτε σήμερα, ούτε σήμερα, ούτε ποτέ. Είμαστε σε μια πολύ βαθιά ύφεση. Η έξοδος θεωρείται ότι είναι οι εξαγωγές. Άκουσα εκπρόσωπο της ΕΚΤ να αναφέρεται στην αύξηση των πορτογαλικών εξαγωγών. Αυτό είναι το είδος της πρωτοβουλίας που απειλεί και τα υποσκάπτει όλα αυτά και μας ανησυχεί πάρα πολύ. Πρόεδρος. Ναι, τη Λος όλη την αγαπάμε. Επιτροπή Βέρνερ Σούλτς. Ποιος θα μιλήσει εκ μέρους Κομισιόν. Έρχομαι από τη ΓΑΜΑ Εμπορίου. Η κριτική είναι ότι όλα αυτά είναι πολύ λίγα. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη τη επιτροπή σα για τα σχόλιά του Πολύ ενδιαφέροντα για μα. Φυσικά, το πρόβλημα έγκυται ότι πρόκειται για το πρώτο τέτοιο εγχείρημα για τις εξαγωγές πιστώσεις. Επομένως, η πρακτική εφαρμογή της διατύπωσης που περιλαμβάνεται στον κανονισμό του 2011 δεν είναι κάτι εύκολο. Σημείωσα ότι πολλοί βουλευτές πιστεύουν ότι δεν αρκούν όλα αυτά, άλλοι φαίνεται να έχουν διαφορετική ερμηνεία. Νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το συζητήσουμε περαιτέρω. Αλλά φυσικά θα πρέπει να λάβουμε και υπόψη ότι τα κράτη-μέλη και πολλά μάλιστα μας είπαν ότι είναι γενναίο αυτό το εγχείρημα για αυτούς, για αυτά και δεν υπάρχει κάποια μορφή διαλόγου από αυτού. Όμως, θα είναι απαραίτητο να κάνουμε αυτό το εγχείρημα για πρώτη φορά και να συναντηθούμε για το πώς θα εφαρμόσουμε τον κοινωνισμό. Και αν μου επιτρέπετε για κάτι τυπικό, Σα έχουμε στείλει το προκαταρκτικό σχέδιο των εκθέσεων αυτών το Δεκέμβρη. Η τελική επίσημη εκδοχή θα σταλεί το συντομότερο. Αλλά ήδη θέλαμε να σας δώσουμε την ευκαιρία να δείτε την ουσία των εκθέσεων των κρατών μελών και να ακούσουμε τα ουσιαστικά σχόλιά σα. Αλλά φυσικά η επίσημη εκδοχή θα ακολουθήσει. Και ισχύει και για την ε, διαπραγματευτική έκθεση. Η Κομισιόν προβλέπει στον κανονισμό 1233 του 2011 όπως εξηγήσαμε και στην επιστολή μας στο Πρόεδρο, σημειώσαμε ότι το πρόβλημα θα ήταν ότι θα έπρεπε να φεθούν εκτός του εγγράφου κάποιες διαπραγματεύσεις Παραδείγματο χάρη με τι Ηνωμένε Πολιτείε που ξεκίνησαν μόλι τον ε, Φεβρουάριο του 2012. Εμεί θα θέλαμε να το συμπεριλάβουμε αυτό στην ε, έκθεση διαπραγματεύσεων. Ένα λεπτό εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Ο στόχος μας είναι να βρούμε έναν τρόπο να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για να ε, υποβάλουν καλύτερα τα στοιχεία για αυτέ τι δραστηριότητε. Είναι ένα πρόβλημα μεθοδολογική φύσεως που θέλουμε με την μήνυα ακρόαση να το εξετάσουμε και θα ήθελα να πω στον αξιότιμο συνάδελφο Ντάρκμουθ ότι, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ε, είναι ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ακόμα υπόκειται σε κάποιο βαθμό στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ότι οι εξωτερικές μας ε, συναλλαγέ πρέπει να είναι υπόλογοι σε σχέση με τι ε, ε, με τις συνθήκες και όσο παραμένετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμορφωθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Την επόμενη φορά η ανταλλαγή απόψεων θα συμπληρωθεί με μία μήνυα ακρόαση που θα λάβει χώρα την επόμενη, στην επόμενη τακτική μας συνεδρίαση στις 28 Μαρτίου. 20 Μαρτίου, συγγνώμη. 20 Μαρτίου είναι η επόμενή μας συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα στη συνεδρίαση.